Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Ξεκινάμε τη σημερινή μας συνεδρίωση και από εδώ και πέρα θα συνεχίσω στα ουγγρικά. Έχουμε λοιπόν το, επόμενο σημείο, το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι η έγκριση της ημερήσιας ε, διάταξης. Την περασμένη Παρασκευή σας ε, στείλαμε την τελευταία εκδοχή της ε, εκδοχής ε, για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Νεολαία 2013-2015. Δεν είχαμε κάποια σχόλια, επομένως εγκρίνεται αυτή η τροποποίηση που έχουμε προτείνει. Διερμηνίαση. Μερά διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες, μεταξύ των οποίων και στα ελληνικά, τα οποία μπορείτε να μιλήσετε και να ακούσετε. Η συνεδρίαση επίσης ε, μεταδίδεται ζωντανά μέσω web streaming. Όσον αφορά τις αποφάσεις της τελευταίας συνεδρίασης των συντονιστών, θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι στη συνεδρίαση της 25ης Απριλίου Έγινε η συνεδρίαση και μετά στις 27 Απριλίου λάβατε τα σχετικά πρακτικά. Δεν υπήρχε κάποια ένσταση ή κάποια αντίρρηση, επομένως εγκρίνονται και τα, οι αποφάσεις των συντονιστών. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία. Έχουμε μια ψηφοφορία για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αύξηση της ποικιλομορφίας της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ε, αγορά κεφαλαίων. Ο κύριος Μόργανο είναι ο εισηγητής, δυστυχώς όμως δεν μπορεί να παραβρεθεί. Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή είναι η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Έχουμε ήδη συζητήσει τη γνωμοδότηση. Στις 26 Απριλίου εξέπνευσε και η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Ε, υπευλήθησαν ε, κάποιες τροπολογίες και έχουμε και έξι συμβαστικές προτάσεις. Μπορούμε να περάσουμε απευθεία στην ψηφοφορία, εκτός και αν θέλει κάποιος να λάβει το λόγο εκ μέρους του συντάκτη της χνομοδότησης, που όπως σας είπα δεν μπορεί να παρευρεθεί. Δεν βλέπω κάποιον, επομένως περνάμε απευθεία στην ψηφοφορία. amendment number... Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. Υπέρ, για τη συμβαστική τροπολογία 3, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 13, υπέρ, κατά, αποχές, Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά να κάνουμε μια επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 12 έχει αποσυρθεί, συγγνώμη. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 31 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά πρέπει να κάνουμε μια επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 33 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Καταπίπτει. Τροπολογία 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίνεται. 48 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε της ψηφοφορίας. 17 υπέρ, κανείς κατά και δύο αποχές εγκρίνεται συγχαρητήρια στο συντάκτη της νομοδότησης. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν παρόντες για την ψηφοφορία και να συνεχίσουμε με την ημερήσια διάταξη. Και τώρα θα ξαναμιλήσω γκρικά. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι ο προπολογισμό του 2017, εντολή για τον τριμερή διάλογο. Η συγητής είναι ο κύριος ε, Σδρογεύσκη. Η Επιτροπή μας καταρτίζει γνωμοδότηση για την Επιτροπή Προϋπολογισμών και ο συντάκτης είναι ο ίδιος με τον ε, προπολογισμό του 2016. Να σας πω ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι αύριο στις 12. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας προβλέπεται για τις 21 Ιουνίου. Κύριε Ζρογεύσκη, να σας δώσω το λόγο. Παρακαλώ. Pani Przewodnicząca, Szanowni e, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να σα ευχαριστήσω όλους θερμά γιατί καταφέραμε για ένα ζήτημα που αφορά προϋπολογισμό να επιτύχουμε μια ευρεία συνένεξη μεταξύ μας. Δεν είναι πάντοτε δηλαδή, δεν συμβαίνει πάντοτε αυτό, αλλά αυτή τη φορά τα καταφέραμε και μάλιστα υποστηρίζουμε τις, ε, και τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Υπάρχει κάποιο θέμα διερμηνίας. Okay? Μπορείτε να μ' ακούσετε, ρωτάει ο κύριος Δρογεύση, μ' ακούτε κανονικά όλοι. Τι teraz, czy teraz... Εντάξει, τώρα υπάρχει διερμηνία. Καλώς, αφού με ακούτε, με ακούτε όλοι καλά, να ξαναρχίσω. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους όσους συμμετείχατε σε αυτή τη συζήτηση, όλους τους συναδέλφους, γιατί συχνά όταν έχουμε να κάνουμε με γνωμοδοτήσεις ε, βέβαια καταφέρουμε να έχουμε μια συνένεση αλλά εδώ παρότι πρόκειται για ένα ζήτημα προπολογισμού έχουμε και υποστήριξη ό,τι αφορά τις τροπολογίες πράγμα βέβαια που καθιστά πολύ εύκολη τη δική μου δουλειά. Ε, σήμερα υπάρχουν μία σειρά από πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία θα επηρεάσουν ε, τον προπολογισμό για το 2017. Αναφέρουμε συγκεκριμένα στη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση αλλά ε, και στην ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου, το Mid-Term review, το επωνομαζόμενο. Όταν έχουμε να κάνουμε εδώ λοιπόν με ζητήματα εκπαίδευσης και γενικά πολιτισμού και παιδείας, ε, τα πράγματα συνήθω δεν είναι τόσο καλά, αλλά εδώ εμείς επιμένουμε για μία ακόμα φορά, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση ειδικότερα του Erasmus Plus. Ε, αναφερόμαστε δηλαδή σε στοιχεία τα οποία δεν έχουν λάβει την κατάλληλη χρηματοδότηση και ότι θα πρέπει να συνεχιστεί και εκείνα τα οποία θέλουμε εμείς ως Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας να προτείνουμε ως δικά μας σχόλια είναι το εξής. Ενισχύουμε τα όσα προτείνονται ήδη, θέλουμε ε, ειδικότερα ε, το Erasmus ε, συν το Erasmus Plus να συνεχιστεί και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να οδηγηθούμε σε μια κατάσταση όπου θα υποχρηματοδοτηθεί αυτό το πρόγραμμα. Μετά. Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης για την Ευρώπη. Είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, όπως και η Ευρώπη για τους πολίτες, το, τα οποία είναι και αυτά πάρα πολύ σημαντικά προγράμματα. Και εγώ κάθε φορά έχω αναφέρει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις Στρατηγικές Επενδύσεις που εντάσσεται ακριβώς στο επωνομαζόμενο σχέδιο Juncker θα πρέπει να λαμβάνει εξίσου υπόψη τα ζητήματα παιδείας. Και δύο ακόμα στοιχεία που θα ήθελα να αναφέρω ως προς τις προτάσεις που κάνουμε. Να πω ότι ήδη από πέρσι είχαμε αναλάβει κάποιες υποχρεώσεις κατά την έγκριση δηλαδή του προηγούμενου σχεδίου του προϋπολογισμού και κατά συνέπεια είναι σημαντικό η πρωτοβουλία την οποία ξεκινήσαμε τότε σε ό,τι αφορά την απασχόληση για τους νέους να τις δώσουμε τη συνέχεια που χρειάζεται. Και κάτι ακόμα σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό και την αξιολόγηση του προπολογισμού από την πλευρά τη Επιτροπή, να πούμε ότι η σχετική διαδικασία έχει παραταθεί κατά έναν συμπληρωματικό μήνα από την πλευρά τη Επιτροπή, δηλαδή την πρόταση του σχεδίου ε, προπολογισμού. Και εμεί, στο επίπεδο των συντονιστών, συμφωνήσαμε από την πλευρά τη δική μα Επιτροπή να προβούμε σε μια συζήτηση, σε μια ανταλλαγή απόψεων ως προς το πώς θα αντιδράσουμε απέναντι σε αυτό. Ε, και ήδη ανέφερε κάτι και η Πρόεδρος, πάντως νομίζω πως στην επόμενη συνεδρίαση θα, ε, έως, ε, θα έχουμε αποφασίσει το ποια προσέγγιση θα ακολουθήσουμε και ε, θα πρέπει κατά συνέπεια μέσα στι επόμενε μέρε να συμφωνήσουμε ω προ τα τελικά στοιχεία που θα περιληφθούν στη δική μα νομοδότηση. Πάντω να πω ότι πραγματικά βλέπω ευρεία υποστήριξη από του συναδέλφου, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τι δικέ μα προτάσει αλλά και προτάσει από υπόλοιπε επιτροπέ. Οπότε δεν νομίζω πω θα υπάρξει κανένα πρόβλημα με την έγκριση εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα έχουμε περίπου 30 λεπτά για ερωτήσεις και απαντήσεις. Σας ακούσουμε λίγο τους και και μετά όποιον συνάδελφο επιθυμεί να μιλήσει παρακαλούμε ενημερώστε μας αν θέλετε να μιλήσετε και όσον αφορά τους και δίνουμε στον καθένα 2 με 3 λεπτά και στους υπόλοιπους ένα με δύο λεπτά. Δεν ζητά να μιλήσει κανείς από τους κοιόδους εισηγητές. Ο κύριος Μαραγκάρ, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι στα αυτά τα θέματα του προπολογισμού πάντα έχουμε την ίδια εντύπωση εκφράζουμε πολύ καλές προθέσεις, ε, την κατάλληλη ορολογία, ε, όλοι πολύ ευγενικά και πολιτισμένα, αλλά όλα αυτά δεν μεταφράζονται σε πρακτικά αποτελέσματα, τουλάχιστον από πλευράς μας, από πλευράς Επιτροπής ε, Πολιτισμού. Πρόκειται βέβαια, για ένα θέμα το οποίο σε μεγάλο βαθμό είναι εκτός Αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, επομένως δεν καλύπτεται και από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό ακριβώς ε, ο ρόλος ο δικό μας ε, και από πλευρά προπολογισμού είναι να προωθήσουμε, να δώσουμε κίνητρα, να καθορίσουμε προγράμματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ε, και θα τα διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι όλα έσα έγιναν από πλευράς ε, εισηγητή είναι σωστά και μπορούμε να συμφωνήσουμε μαζί του και σίγουρα στις μέρες που έχουμε στη διάθεσή μας για να εργαστούμε και να ε, καταλήξουμε σε συμβαστικές ε, προτάσεις, ελπίζω ότι θα έχουμε και το επίπεδο συμφωνίας που χρειάζονται και να καταλήξουμε σε μια συνένεση. Θα ήθελα να σταθώ σε κάποια πολύ συγκεκριμένα προγράμματα ε, τα οποία όταν θα συζητήσουμε στις τροπολογίες θα μπορέσουμε ίσως να τα συζητήσουμε και με την πάσα λεπτομέρεια. Πρώτον, εξακολουθεί να υπάρχει ένα πρόβλημα στις πληρωμές, όχι μόνο από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από πλευράς κρατών μελών. Και θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η ευθύνη αυτή ε, μπορεί να οδηγήσει και σε αρνητικές συνέπειες, όπως γίνεται πάντα με την ανεπαρκή διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδύλιων. Δεύτερον, ε, στα πλαίσια του Erasmus Plus, που σίγουρα είναι το πρώτο και πιο σημαντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα και αυτή τη στιγμή είναι και από τα λίγα τα οποία εξακολουθούν να διατηρούν το γόητρο και την θετική εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αλλά χρειάζεται διεύρυνση, χρειάζεται ενίσχυση και χρειάζονται και κάποιοι νέοι προσανατολισμοί οι οποίοι αδιαφυσβήτητα θα έχουν και συνέπειες για τον προπολογισμό. Εμείς κάνουμε κάποιες προτάσεις. Εμείς καταρχάς ε, προτείνουμε ενίσχυση ε, του γραμμής προϋπολογισμού για την επαγγελματική κινητικότητα. Μας φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε σε τόσο μεγάλο ποσοστό αν νεανικής ανεργίας και εγκατάλειψης των σχολείου, από αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να μην υπάρχει κανένα όριο στις προσπάθειες που πρέπει να γίνουν για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στον τομέα αυτό. Επίσης, εδώ Προφανώς τα προγράμματα τα οποία απευθύνονται σε μικρά έργα και στο ρόλο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και κοινωνικών οργανώσεων πολύ δύσκολα μπορούν να υλοποιηθούν στα πλαίσια του Erasmus+. Αυτό πρέπει να γίνεται σε, συντονιστό, ε, σε συντονισμό με τις εθνικές υπηρεσίες, οι οποίες είναι τόσο εθνικές και είναι τόσες πολλές οι υπηρεσίες που σημαίνει ότι δεν μπορούν να επιδείξουν την κατάλληλη ευελιξία για να υλοποιηθούν αυτά τα προγράμματα και είναι απαραίτητο να έχουμε αυτούς τους συνομιλητές. Επίσης, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι και το έχουμε συζητήσει επανειλημμένως ότι πρέπει ε, να υπάρχει και μία γραμμή απλοποίησης να αλλάξουν λίγο οι διαδικασίες ε, ώστε τα προγράμματα του Erasmus Plus ε, να προχωρούν πιο γρήγορα, πιο εύκολα και να μπορούν να απορριφήσουν στο 100% τα όσα ε, προβλέπονται από τον προϋπολογισμό. Και τέλος, για να μην μακρηγορήσω και πάρα πολύ, νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να επενθυμίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών ε, Επενδύσεων μας χρωστάει ε, και αυτό το χρέος ε, δεν έχει ακόμα αποπληρωθεί, επομένως πρέπει να δοθούν αυτά τα κονδύλια, πρέπει κάπως να βρεθούν αυτά τα κονδύλια που χάθηκαν στην αρχή και Επίσης, ε, αλλάξανε τα πράγματα και στο Εράσμους, μας το εξήγησαν και κάποιοι κοινωνικοί εταίροι. Κάποιες από τις γραμμές ε, είτε δεν απορροφούνται καθόλου ή δεν ε, χρησιμοποιούνται όλα τα κονδύλια. Παραδείγματο χάρη οι γραμμές δανεισμού του Εράσμους. Θα πρέπει λοιπόν να προβλέψουμε με μεγαλύτερη ευελιξία, καλύτερη διαχείριση αυτών των δανειοδοτήσεων είναι δανειοδοτήσει, οι οποίες έχουν πολύ σημαντική δυνατότητα εντός του ράσμους και τελικά δεν χρησιμοποιούνται γιατί δεν έγινε κατάλληλη διαχείριση και δεν εφαρμόστηκαν καταλήλω. Επομένω. Ή θα φροντίσουμε να απορροφάτε το 100% ή το πιο λογικό να προβλέψουμε μηχανισμούς εσωτερικής ευελιξίας εντός του Εράσμους ώστε να μπορούν να διατεθούν τα κονδύλια και να δίνονται χρήματα σε προγράμματα τα οποία έχουν ελλείψεις ε, και να παίρνουμε τα χρήματα από κάποια άλλα στα οποία υποτίθεται ότι υπάρχουν άλλες προβλέψεις. Υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα τα οποία είναι ίσονος σημασίας, είναι πιο συγκεκριμένα και επομένως ε, θα δούμε για παράδειγμα και τι γίνεται με το Youth Guarantee, την εγγύηση για την νεολαία, το οποίο δεν χρειάζεται μόνο ε, κονδύλια, αλλά χρειάζεται να επιδείξει και αξιοσύνη η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει να καλύψει τους αρχικούς της στόχους αυτό το πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Κάποιος άλλος που θα ήθελε το λόγο από τους και ο ο κ. Κουντής, παράδειγμα. Όχι. Όχι. Να δώσω το λόγο στη συνάδελφη την κυρία Σόντροβα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας για την γνωμοδότηση αυτή, ε, η οποία θεωρώ ότι αναφέρει όλα τα σημαντικά χρηματοοικονομικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας και τα οποία διασφαλίζουμε και εμείς ε, στο πλαίσιο της Επιτροπής μας. Τις τελευταίες ημέρες ε, στην ε, επίσκεψη στην Κολονία είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε ότι το Erasmus Plus είναι ένα σημαντικό και χρήσιμο εργαλείο το οποίο χαίρει ιδιαίτερη εκτίμηση στα σχολεία, στι μη κυβερνητικέ οργανώσει και σε όλου του πολίτε. Το υποστηρίζουμε λοιπόν και υποστηρίζουμε και τα χρηματοοικονομικά μέσα για το Erasmus Plus. Επίση έχουμε και προτεραιότητε αυτή τη στιγμή όπως για παράδειγμα για τους νεαρούς πρόσφυγες, νεαρούς μετανάστες, για την κοινωνική ένταξη των νέων και ούτω καθεξής. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε την γνωμοδότηση αυτή. Θα ήθελα να τονίσω και κάποιες άλλες προτεραιότητες που αναμένουμε να δούμε το 2017 υπάρχουν ε, αυτές οι προτεραιότητε 2017 και άλλε φυσικά και εγώ θα υποστηρίξω αυτή την γνωμοδότηση. Θέλω να πω ευχαριστούμε εκ μέρους τη Επιτροπή. Θα ήθελε κάποιο να παρέμβει. Κάποιος εκπρόσωπο τη επιτροπή. Όχι, όπως φαίνεται. Ωραία, ευχαριστούμε. Μπορούμε να κλείσουμε αυτό το σημείο το πρώτο σημείο συζήτησης. Α, ε, θέλει ξανά να πάρει το λόγο ο Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να προσθέσω κάτι για όσα είπε ο κύριος ε, Μαραγκάλα. Είναι πολύ σημαντικό να διορθωθεί το πρόβλημα προς τους δικαιούχους από τα προγράμματα που υπάρχουν. Εγώ στη φάση της γνωμοδότησης θα προσπαθήσω να συμπεριλάβω αυτή την παρατήρηση γιατί είναι σημαντική. Θα ήθελα να σημειώσω ότι έχουμε μια άριστη πρόταση για το επόμενο έτος. ώστε να μειωθούν ε, ή ε, ε, ε, κάποιες δεσμεύσεις για αυτά τα προγράμματα είναι σημαντικό γιατί πρέπει να δούμε αναλογικά τι γίνεται σε σχέση με τα άλλα προγράμματα. Ένα δεύτερο πράγμα που θα ήθελα να σας υπενθυμίσω είναι η πολύ σημαντική σωστή πολιτική πληροφοριών και επικοινωνίας. Αυτό αντεποκρίνεται και στις επιθυμίες που έχουν εκφραστεί εδώ. Έτσι λοιπόν έχω συμπεριλάβει μαζί με το Erasmus Plus και άλλες πολιτικές ε, για την πολιτική ε, παιδείας ε, ώστε να βελτιωθεί και να βελτιωθούν και τα όσα κάνουμε εμείς και τα όσα κάνουν τα κράτη-μέλη. Οπότε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για αυτή την ομοδότηση. Ευχαριστούμε. Μπορούμε τώρα πραγματικά να κλείσουμε το σημείο αυτό. Ζητώ συγγνώμη που δεν σας έδωσα το λόγο για την απάντηση. Περνάμε στο σημείο 6. Η Ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δυνατότητε και προκλήσει. Ε, η συγκήτρια, η συνάδελφο κυρία Αντινόλφη. Ε, η γνωμοδότηση αυτή αναφέρεται στις ε, αρνητικέ επιπτώσει για τα κοινοβούλια λόγω ε, του όλο και μικρότερου ενδιαφέροντο εκ μέρου των πολιτών στις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης, της οικονομικής κρίσης και εκφράζεται η ανάγκη να ανανεωθεί κατά κάποιο τρόπο η σχέση των πολιτικών και του, των λαών ε, και στο πλαίσιο της πολιτικής διαδικασίας ε, και να επανακαθοριστεί ο ρόλος των πολιτικών κομμάτων για την καταπολέμηση της ε, διαφθοράς. Έτσι λοιπόν τα διάφορα ψηφιακά εργαλεία και οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες μπορούν να αποτελέσουν μια δημιουργική λύση για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στο δημοκρατικό σύστημα, ειδικότερα μεταξύ των νέων. Η Επιτροπή ΑΦΚΟ, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, θα υποβάλει στις 30 Ιουνίου την έκθεση πρωτοβουλίας και μετά από μια ανταλλαγή απόψεων η δική μας σκιώδηση ε, για την Επιτροπή Κάλτε είναι η κυρία Ντινόλφη. Εμείς ε, της αναθέσαμε αυτό το ζήτημα λόγω των γνώσεων που έχει στο ζήτημα της ηθαγένειας. Πριν της δώσω το λόγο, θα ήθελα να επενθυμίσω είναι ότι η υποβολή τροπολογιών μπορεί να γίνει μέχρι την Τετάρτη 7 Ιουνίου στις 3 το μεσημέρι. Ψηφοφορία στην Επιτροπή μας θα λάβει χώρα στις 12 Ιουλίου. Κύριε Αντινόρφη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Κατά την άποψή μου, για μένα ήταν τιμή το να οριστώ συντάκτρια από τη συνεδρία των συντονιστών και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό η Επιτροπή μας, η Επιτροπή Πολιτισμού δηλαδή, να ε, ε ακουστεί ως άποψη για ένα τόσο σημαντικό θέμα ώστε να εντάξουμε, να συμπεριλαβηθεί και στην έκθεση και η δική μας άποψη, η άποψη της Επιτροπής μας όσον αφορά την Ιθαγένεια. πέραν των όσων φυσικά θα γράψει η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Το θέμα είναι ότι τα νέα μέσα και οι νέες τεχνολογίες έχουν καθορίσει και ακόμα καθορίζουν σοβαρές ε, μεταβολές ε, τόσο όσον αφορά τους τρόπους εκμάθησης ε, όσο και τη διάδοση των νέων πληροφοριών. Έτσι λοιπόν με αυτά τα νέα τεχνολογικά μέσα αλλάζουν τα πράγματα και όσον αφορά την ηθαγένεια και αλλάζει και ο τρόπος ε, συμμετοχής στην πολιτική ζωή. Έχει αλλάξει η έννοια της δημοκρατίας κατά την απόψή μου και εμείς πρέπει να έχουμε συνείδηση αυτού του γεγονότος, κυρίως επειδή είμαστε συνομοθέτες. Οι πολίτες παλιότερα κάθε πέντε χρόνια απλά πήγαιναν να ψηφίσουν. Και μετά υπήρχε ένα κενό μεταξύ των δύο εκλογών, εκλογικών περιόδων, ενώ αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή. Πολύ πιο εκτενή. με αυτό το εργαλείο, με το smartphone, με τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα. Οι πολίτε ουσιαστικά ανά πάσα στιγμή μπορούν να συμμετάσχουν και καθημερινά στην ε, ζωή μας, στη ζωή των θεσμικών οργάνων. Γι' αυτό τον λόγο πιστεύω ότι η αντιπροσωπευτική δημοκρατία πρέπει να ενισχυθεί και να πλησιωθεί από τέτοια εργαλεία άμεσης δημοκρατίας ε, που διευκολύνεται σήμερα λόγω των νέων μέσων και των νέων τεχνολογιών. Ο νομοθέτης πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσει τις αλλαγές, ε, να τις ελέγχει, να τις διαχειρίζεται, ώστε να βεβαιώνεται ότι τα νέα αυτά μέσα χρησιμοποιούνται υπέρ της δημοκρατίας, υπέρ των πιο αδυνάμων, των περιθωριοποιημένων και όχι μόνο για τη διατήρηση του status quo, των λόμπι ή των επιχειρηματικών συμφερόντων. Εμείς ως μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού θεωρώ ότι έχουμε το καθήκον να ε, εντοπίσουμε τους πιθανούς κινδύνους και τα πλεονεκτήματα αυτών των μεταλλαγών, ώστε, αντιμετωπίζοντας τα διάφορα ζητήματα που ε, ναι, έτσι τα διάφορα ζητήματα που παρουσιάζονται με τα δια, ε, διάφορους τρόπους ε, εκμάθησης που προσφέρουν τα νέα μέσα μπορούμε να ευνοήσουμε μία εκμάθηση πιο συγκεκριμένη και με πιο κριτικό πνεύμα ε, σε κάθε είδους αυτή η χρήση των νέων μέσων πρέπει να ανοιχτεί διαφανεί όσο δυνατόν περισσότερο οριζόντια, ώστε να διασφαλίζει την ανεξαρτησία και να αποφεύγεται οποιαδήποτε χειραγώγηση μέσω αυτών των πληροφοριών. Ε, χρειαζόμαστε και συγκεκριμένες προσπάθειες για να ευνοήσουμε τη νέα ε, ψηφιακή συμμετοχή των πολιτών στο πολιτικά δρόμενα προσφέροντας και μεγαλύτερο χώρο. Το δικό μας πολιτικό κίνημα ανέκαθεν χρησιμοποιούσε πλατφόρμες τέτοιου τύπου και τώρα χρησιμοποιεί μια νέα πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τους εκπροσώπους ε, στα θεσμικά όργανα και συμμετοχής ε, στην προετοιμασία των πράξεων. Έτσι λοιπόν ε, σημειώνω ε, με μεγάλη μου χαρά ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται μπροστά με αυτού του είδου του πειραματισμού. Πράγματι, το Κοινοβούλιο έχει ξεκινήσει ένα πιλωτικό έργο τέτοιου τύπου που πιστεύω θα πρέπει να προωθηθεί, να ενισχυθεί και να υλοποιηθεί ε, το συντομότερο δυνατόν. Είμαι πεπισμένη ότι ε, έχει οριμάσει η κοινωνία για τη χρήση τέτοιων μέσων, οπότε τα έργα αυτά θα πρέπει να τα να τα χρησιμοποιούμε έτσι ώστε ε, να μπορούν να αξιολογηθούν, να βελτιωθούν, να, αξιολογηθούν οι πιθανοί κίνδυνοι και να προωθηθούν οι θετικές πτυχές. Δύο ε, θέματα δεν πρέπει να ξεχνάμε κάνοντας την ανάλυση αυτή. Πρώτον, στο ψηφιακό, το ψηφιακό χάσμα, ε, τόσο όσον αφορά τις υπεδομές, όσο και το πολιτιστικό χάσμα. Και δεύτερον, την ψηφιακή ένταξη Πιστεύω ότι τα δύο αυτά ζητήματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν πολύ συγκεκριμένα και πολύ σωστά, ώστε να καταλήξουμε σε ε, λύσεις και σε ψηφίσματα αποτελεσματικές ε, και ταχείες ε, παρέχοντας έτσι πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλους τους πολίτες να το θεωρήσουμε αυτή την πρόσβαση ένα θεμελιώδες δικαίωμα που θα φυλάσσεται από το Σύνταγμα για παράδειγμα στην Εστονία υπάρχει ένα συνταγματικό δικαίωμα πρόσβαση στο διαδίκτυο Θεωρώ επίσης ότι όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν το δικαίωμα πρόσβαση στο δίκτυο όχι μόνο να έχουν επαρκή ψηφιακή παιδεία ώστε να εξομαλυνθούν οι κοινωνικές και οικονομικές ε, ανισότητες αλλά για να προστατεύσουμε και την ισότητα και την ελευθερία και την πολιτική, δημοκρατική συμμετοχή στην πολιτική ζωή. Συγκεκριμένα προγράμματα λοιπόν εκπαίδευση θα πρέπει να δημιουργηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα εστιάζονται και θα προορίζονται κυρίως για τις μειονεκτούσες κατηγορίες ε, για τις ε, πολιτών ε, όπως είναι ας πούμε οι πολιτές με θα ήθελα να πω ότι στο σχέδιο αυτό κειμένου έχω υπογραμμίσει τα σημαντικότερα σημεία που δεν αποτελούν παρά μια αφετηρία φυσικά διότι υπάρχουν και περιορισμοί φυσικά ε, στο πόσο μεγάλο μπορεί να είναι το κείμενο. Θέλω να πω ότι στις διάφορες επαφές που θα έχουμε θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε ένα ικανοποιητικό κείμενο το οποίο να αντικατοπτρίζει και να αποτυπώνει τις διάφορες θέσεις και ευαισθησίες ε, εντό της Επιτροπής Πολιτισμού. Από πλευράς μου μπορώ να σας πω ότι εγώ δεσμεύομαι προς αυτή την κατεύθυνση και είμαι πεπισμένη ότι πρέπει οπωσδήποτε να προωθήσουμε την άποψη της Επιτροπής μας όσον αφορά τα θέματα ηθαγένειας, ώστε αυτό να είναι απόλυτα σαφές στην έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχουμε γύρω στα 30 λεπτά τώρα στη διάθεσή μα ε, για τη συζήτηση σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Καταρχήν θα δώσουμε το λόγο στους σκιώδες εισηγητέ και μετά στους υπόλοιπου συναδέλφους που θέλουν να πάρουν το λόγο. κυρία Φεχάν, λοιπόν, ε, καταρχήν. Ε, ευχαριστώ πριν το λόγο εκ μέρου του σκιώδου συγκεκριτή Σφαίρ, γιατί δεν κατάφερα να παρευρεθεί σήμερα εδώ γιατί υπάρχει μια ε, πολιτική συνάντηση για την 40η ε, επέτειο της δημιουργία του ΕΛΚ στο Λουξεμβούργο σήμερα. Και αυτό αποτελεί την ε, αιτία για την οποία πολλά μέλη του ΕΛΚ δεν παρευρίσκονται σήμερα εδώ, αλλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι χρειάστηκαν να μεταβούν σε άλλε επιτροπέ για να του αντικαταστήσουν. Η κυρία Φέρ, λοιπόν, τόνισε επανειλημμένα ε, το, την ανάγκη του να σταματήσουμε την μείωση της δημοκρατικής συμμετοχής ε, των ε, πολιτών την οποία έχουμε παρατηρήσει κατά τι τελευταίε δύο δεκαετίε. Ε, άρα λοιπόν η άμεση δημοκρατία και η ηλεκτρονική δημοκρατία αποτελούν εργαλεία μέσω των οποίων μπορούμε να προσελκύσουμε περισσότερο του ανθρώπου, ειδικότερα του ε, νέου, για τη συμμετοχή του, την αυξημένη συμμετοχή του στι δημοκρατικέ ε, διαδικασίε και κατά συνέπεια να μειώσουμε το δημοκρατικό έλλειμμα. Αλλά υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματο. Δηλαδή υπάρχουν κάποιε παγίδε στην αυτήν την άμεση δημοκρατία σε σύγκριση με την αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Οπότε η άμεση δημοκρατία στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν είναι καλά ενημερωμένοι οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, γιατί κάτι τέτοιο βέβαια μπορεί να οδηγήσει στο να ε, χειραγωγούνται από την ε, προπαγάνδα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει κατάλληλη ενημέρωση, ειδικότερα των νέων, τους, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους στο πλαίσιο των δημοκρατικών διαδικασιών με καλό τρόπο. Θεωρούμε, θεωρεί συνάδελφος ότι είναι καλά διατυπωμένη η γνωμοδότηση, αλλά θα μπορούσαν να βελτιωθούν οι παράγραφοι 3 και 4. Ειδικότερα χρήση της λέξης critical δεν είναι τόσο ενδεδειγμένη, θα μπορούσαμε να λέμε proper knowledge, κατάλληλη γνώση δηλαδή τη Ευρωπαϊκή Ένωση και επίση θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη έμφαση στον θετικό ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην παράγραφο 5 γίνεται λόγο για decentralized sources, δηλαδή αποκεντρωμένε πηγέ ε, πληροφοριών. Ε, θα πρέπει να αναδιατυπωθεί αυτό το σημείο και να λέμε ότι αυτές οι αποκεντρωμένες ε, ε, πηγές πληροφοριών όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην δίνουν απευθείας ε, απαντήσεις. Επίσης, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον την ελλειπή ε, γνώση των ε, δημοκρατικών ζητημάτων. Ε, να πούμε ότι σήμερα οι πολίτε συχνά δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν ποιε είναι αξιόπιστε και λιγότερο αξιόπιστε πηγέ πληροφοριών. Επίση, κάτι ακόμα που θα πρέπει να αναφερθεί από την κυρία Τινόλφη είναι η πρόσβαση στο διαδίκτυο από την πλευρά όλων, ώστε να μειωθεί και το ψηφιακό χάσμα. Επίση, η ηλεκτρονική δημοκρατία είναι πολύ σημαντική και στο πλαίσιο του σημερινού ευρωσκεπτικισμού, ακριβώ επειδή θα μπορούσε να ε, έχει επιπτώσει σε ό,τι αφορά την αίσθηση του, του ανήκειν των ε, πολιτών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώ εκεί βρίσκεται και ο κίνδυνο του να βρεθούν θύματα προπαγάνδα οι Ευρωπαίοι πολίτε. Ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο συνάδελφο που θα ήθελε να πάρει το λόγο από του Κιώδη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετική δουλειά που έκανε. Πραγματικά πρόκειται για ένα πολύ καλό σχέδιο γνωμοδότηση. Ε, να πω και ότι συμμερίζομαι τον ενθουσιασμό της εισηγήτριας ε, για αυτό το ζήτημα. Ε, επίσης, ε, μου αρέσει το γεγονός ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη γνωμοδότηση, στην συμμετοχή στα κοινά και ειδικότερα στην ψηφιακή συμμετοχή, δηλαδή την άρση των περιορισμών. Αλλά βέβαια εδώ το ζητούμενο για την ηλεκτρονική δημοκρατία δεν είναι μόνο να υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία στη διάθεση των πολιτών, αλλά να αλλάξουν και νοοτροπίε, ούτω ώστε δηλαδή οι πολίτε να μην είναι απλά καταναλωτέ σε ψηφιακή, αλλά πραγματικά ενεργοί πολίτε στο πλαίσιο διασυνδεδεμένων κοινωνιών. Ε, και εγώ, καθώ ε, κατάγομαι από την βορειοδυτική Αγγλία, ε, προέρχομαι από μία από τι ε, ε, πλέον διασυνδεδεμένε πόλει του κόσμου, το Μάντσεστερ. Οπότε πραγματικά αυτό το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό για μένα από εκεί όπου κατάγομαι. Όμω, από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί να υπάρξει ηλεκτρονική δημοκρατία αν δεν υπάρχει συμμετοχή, ένταξη δηλαδή ενεργό συμμετοχή ειδικότερα των ευάλωτων ομάδων. Οπότε συμφωνώ με αυτή την ε, προσέγγιση τη ηγετρία. Πάντω, ε, στο πλαίσιο των τροπολογιών θα ήθελα να προτείνω το να δώσουμε περισσότερη έμφαση σε ορισμένα στοιχεία. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το να εκπαιδεύσουμε ε, του ε, δασκάλου και του άλλου εκπαιδευτέ, σε ό,τι αφορά την χρήση των τεχνολογιών τη πληροφορία και των επικοινωνιών, όταν οι ίδιοι αυτοί εκπαιδευτέ και δάσκαλοι δεν νιώθουν άνετα με τέτοιου είδου τεχνολογίε, αλλά καλούνται να προετοιμάσουν μια νέα γενιά ανθρώπων οι οποίοι θα ζουν σε έναν νέο ε, τελείως διαφορετικό κόσμο τον οποίο ακόμα δεν μπορούμε να φανταστούμε. Οπότε ε, θα πρέπει να, έχουν, ε, να τους δώσουμε τις κατάλληλες δεξιότητες και τις τις κατάλληλε γνώσει για τη διδασκαλία. Η αδερφή μου είναι δασκάλα και ε, πέρα από όλα, όσα είναι υποχρεωμένη να κάνει θα πρέπει τώρα ε, να, είναι, να αναλάβει τον ρόλο κάποιου ο οποίος προωθεί ε, τον ψηφιακό κόσμο αλλά χωρίς να έχει λάβει καμία περαιτέρω καθοδήγηση, καμία σχετική εκπαίδευση. Οπότε θα πρέπει να διατεθούν οι κατάλληλοι πόροι από την πλάτη των κρατών μελών προς τους εκπαιδευτές. Επίσης, οι προκλήσεις αλλά και οι δυνατότητες ε, που, δίνει, ε, που δίνουν σχετικές ε, τεχνολογίες για την πολιτισμική ποικιλομορφία. Εδώ πράγματι μπορούν να δημιουργηθούν νέες πλατφόρμες ώστε να υπάρξουν να υπάρξει και καλύτερη πρόσβαση των όσων δημιουργούν σε, ε, μεγαλύτερους, ε, σε μεγαλύτερα κοινά, αλλά υπάρχουν εδώ και κάποιοι μεγάλοι παίκτε εντό εισαγωγικών οι οποίοι μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτά τα εργαλεία. Οπότε θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και επίση θα πρέπει να δώσουμε ένα ερέθισμα για να υπάρχει περισσότερη πολιτισμική περιέργεια, αν θέλετε, ε, ούτω ώστε ακριβώ να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το σχετικό δυναμικό. Και εδώ βέβαια πάλι έχουμε να κάνουμε τι σχετικέ τεχνολογίε. Επίση, να αναφερθώ λίγο και στη διάσταση εδώ του φίλου η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και επίσης Εκείνο που θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω είναι οι περισσότερες ανεξάρτητες και ποιοτικέ πηγές πληροφοριών, ούτως ώστε να αξιοποιήσουμε αυτό που μας προσφέρει η ηλεκτρονική δημοκρατία, δηλαδή περισσότερες, περισσότεροι τρόποι ενεργού συμμετοχή. Κατά τη δική μου γνώμη, λοιπόν, οι τρεις πυλώνες θα πρέπει να είναι η ένταξη, η εκπαίδευση και Άρα λοιπόν ε, κλείνοντας να πω ότι είναι πραγματικά μια, ένα ε, πάρα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα, μια πάρα πολύ καλή γνωμοδότηση και αναμένω με ενδιαφέρον και τις μελλοντικέ μας ε, συζητήσεις για αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you, Madam Chairman. Well, some of the, uh, some of the lines... Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το ECR καλωσορίζει την πρόταση αυτή και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε ότι η άμεση δημοκρατία είναι ο μόνος ε, τρόπος για μια δημοκρατική διαδικασία. Τα όσα είπε η κυρία Φερχόιεν για την αντιπροσωπευτική δημοκρατία νομίζω ότι συνάδουν και με τις δικές μας τις απόψεις του θέματος. Καλό είναι από καιρού καιρού να έχουμε και άμεση δημοκρατία υπό τη μορφή δημοψηφισμάτων, αλλά αυτό κυρίω θα πρέπει να επιφυλάσσεται για εκχώρηση κυριαρχία, ε, ε, θέματα σε αυτά το επίπεδα και όχι τα καθημερινά ζητήματα, γιατί ουσιαστικά θα χαθεί η σημασία της ε, εκπροσώπησης ε, οι ε, ε, αιρετοί είναι αυτοί που πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις και μετά ο λαός να κρίνει τις αποφάσεις τους. Ε, να μην έχουμε μια τόσο απλοϊκή εικόνα της άμεσης δημοκρατίας όσον αφορά το να συμπεριλάβουμε τέτοιες αναφορές στα συντάγματα. Η τεχνολογία κινείται πάρα πολύ γρήγορα και εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι τα ε, συντάγματα επηρεάζονται αντιστρόφως ανάλογα με την έκτασή τους. Επομένως θα πρέπει ε, να φροντίσουμε να υποστηρίξουμε ανθρώπους που χρειάζονται υψηλό επίπεδο ψηφιακή πρόσβασης αλλά και ψηφιακέ δεξιότητε. Αυτό έρχεται να ε, προσθεθεί σε αυτά που μόλις είπε η Τζούλη. Δεν θέλουμε απλώς να έχουμε πρόσβαση στον ψηφιακό κόσμο. Πρέπει να υπάρχει και κατάλληλο μορφωτικό υπόβαθρο το οποίο θα επιτρέψει στους πολίτες να κάνουν συνειδητές αποφάσεις ε, ε, διότι αυτή τη στιγμή η ε, πληροφορία και η τεχνολογία της πληροφορικής ε, δεν είναι μόνο θέμα το οποίο πρέπει να διδάσκεται στο σχολείο, είναι θέμα το οποίο καλύπτει οριζόντια όλα τα επαγγέλματα και ακόμα και επαγγελματική κατάρτιση λοιπόν θα πρέπει να γίνεται. Το ECR υποστηρίζει κάποιες από τις προτάσεις της εισηγήτριας και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε και επικοδομητική συνεισφορά όσο προχωρά η πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μαραγκάλ τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Αντινόλφη έλεγε ότι ήταν τιμή για αυτή να μπορέσει να είναι συντάκτρια αυτής της γνωμοδότησης. Εγώ ζηλεύω και λίγο γιατί έχετε δίκιο. Χαίρομαι που είστε εσείς ε, η αρμόδια και που μας υποβάλλετε αυτή τη γνωμοδότηση ακριβώς με τον τρόπο που μας την έχετε υποβάλει. το μόνο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι προτείνει, ότι δίνει κίνητρα, ότι προωθεί ε, τις προσθήκες ε, και τις αλλαγές. Ε, νομίζω ότι όσα λέει εδώ είναι απόλυτα σωστά, τα συμμερίζομαι και εγώ και θα ήθελα ε, πολύ σύντομα να προσθέσω κάτι με το οποίο ελπίζω να συμφωνήσει. Ελοχεύει ο κίνδυνος να χαθούμε σε μια θεωρητική συζήτηση για τα e-tools και να ξεχάσουμε το περιεχόμενο. Διότι προφανώς, δεν είναι αυτό θεωρία, ε, προφανώς αυτή τη στιγμή ο κίνδυνος έλλειψης ισορροπίας μεταξύ της ισχύω των μέσων, της τεχνολογίας, ε, της πληροφορικής και της επικοινωνίας πιο συγκεκριμένα και της περιπλοκότητας του μηνύματος που πρέπει να περιλαμβάνεται ε, μπορεί να είναι πολύ μεγάλες και μπορεί να υπάρχουν και απόπειρα χειραγώγησης, ε, στρέβλωσης και η δημοκρατία, η δημοκρατική συζήτηση σημαίνει να γνωρίζω, να κατανοώ και να αποφασίζω. Άρα, αυτό το οποίο πρέπει να απαιτούμε όταν αναφερόμαστε για παράδειγμα στη γενικευμένη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής, είναι ότι υπάρχει μια προϋπόθεση για να γίνει αυτό. Πρέπει να καλύπτονται λοιπόν και τα τρία θέματα και τα τρία ρήματα. Μαθαίνω, κατανοώ και αποφασίζω. Πρέπει να υπάρχουν γνώσεις, πρέπει να βοηθούν προς την κατανόηση και πρέπει να επιτρέπουν να λαμβάνουμε αποφάσεις. Ιδάλλως θα πάμε στην εντελώ αντίθετη κατεύθυνση. Γι' αυτό ακριβώ και φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικό να προσθέσουμε εδώ και δύο λόγια για την ε, τη δράση, την ενεργό δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, όχι μόνο για να διευκολύνουμε την πρόσβαση, όχι μόνο για να επιτρέψουμε στους πολίτες να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις τεχνολογίες κατά τη δημοκρατική μα συζήτηση, αλλά να είμαστε και ε, υπόδειγμα για αυτή την ενεργό δράση, ε, το σεβασμό της περιπλοκότητας, την κατάλληλη άρτια γνώση των θεμάτων και νομίζω ότι η Επιτροπή μα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα από όσα γίνονται για να επιτρέψει να γίνει συζήτηση εκ παραλλήλου με του πολίτε για τη δική μα τη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Και αυτό ε, γιατί να μην το απαιτήσουμε. Ε, γιατί ε, για παράδειγμα στη συζήτηση για τον προπολογισμό, στην οποία συμμετέχω κι εγώ δεν έχει συζήτηση για να τη δουν οι πολίτες ε, τι γίνεται με τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσε όμως με βάση αυτό να γίνει. Η συζήτηση για την ε, προσφυγική κρίση. Φυσικά είναι ανύπαρκτη συζήτηση γιατί εμείς ως κοινοβούλοι δεν μπορούμε να αποφασίσουμε. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα μέσο, υπάρχει χρήση τη τεχνολογία των πληροφοριών που μας επιτρέπει να έχουμε στοιχεία, αριθμητικά στοιχεία, σημεία αναφοράς ε, και να έχουμε αντικειμενικά μια εικόνα της πραγματικότητας. Πρόσβαση δηλαδή στη δημόσια ζωή και να έχουμε ε, και μεγαλύτερο επίπεδο φιλοδοξίας της δημοκρατικής χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής. Ε, είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι θα τα καταφέρουμε να συμφωνήσουμε και θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε αυτή τη γνωμοδότηση. Δεν ξέρω αν έχει νόημα, ίσως δεν έχει, να υπενθυμίσουμε και τη δυνατότητα η ψηφοφορία στις ευρωπαϊκές εκλογές ε, να γίνεται και με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Μπορεί ίσως να μην είναι ε, δική μας ε, υπόθεση, να μην είναι θέμα Επιτροπής Πολιτισμού ή όχι μόνον Επιτροπής Πολιτισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μαλτέζε. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, ε, να συγχαρώ την Ιζαμπέλα την γιατί έκανε εξαιρετική δουλειά. Πρόκειται για μια ισορροπημένη γνωμοδότηση και νομίζω ότι έχει εξετάσει βάθος ε, και τους λόγους ε, και νομίζω ότι χαίρομαι που ε, ασχολείται κάποιος με τη γνωμοδότηση αυτή από το κίνημα των πέντε αστέρων. Εγώ δεν συμμετέχω σε αυτό το κίνημα, αλλά νομίζω ότι είναι το κίνημα το οποίο μπόρεσε να χρησιμοποιήσει καλύτερα τις νέες μορφές επικοινωνίας στην πολιτική επικοινωνία. Πέραν αυτού, καταρχάς να πω ότι εκτιμώ το γεγονός ότι επισημενονται τα κοινωνικά ζητήματα τα οποία υφέρπουν ε, ε, ενώπιον αυτού του δημοκρατικού αποκλεισμού. Και νομίζω ότι η μικρότερη πολιτική συμμετοχή αυτές τις ε, δεκαετίες συμβαδίζει και με τον αποκλεισμό από την κοινωνία όλο ένα και πιο σημαντικών τμήματων της κοινωνίας. Οι κοινωνικές διαφορές αμβλήνθηκαν, οι οικονομικές και κοινωνικές διαφορές αμβλήνθηκαν και εντός των χωρών και μεταξύ των χωρών. Δεν καταλαβαίνουμε καλά ε, γιατί αυτός που νιώθει περιοθεωριοποιημένος και αποκλεισμένος ε, κοινωνικά και οικονομικά θα πρέπει στη συνέχεια να συμμετέχει περισσότερο στο δημοκρατικό βίο. Και επομένως, ε, από αυτή την άποψη, η Ένωση δεν λειτουργήσε. Δημιούργησε περισσότερες διαιρέσεις και ο στόχος ήταν να δημιουργήσει μεγαλύτερη ισότητα. Μία από τις ε, πηγές ε, διχασμού είναι η πρόσβαση στη γνώση. Η πρόσβαση στα, μέσα, ε, στα νέα μέσα επικοινωνίας και τεχνολογίας. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να ενθαρρύνουμε αυτά τα προγράμματα και είναι και εξίσου σημαντικό να κατανοήσουμε σε τι έχουμε πρόσβαση. Διότι ένα μειονέκτημα του νέου κόσμου της τεχνολογίας, αν υπάρχει, και εγώ σας το λέω ως άνθρωπος που όλη μου τη ζωή δημοσιογράφος ήμουν, είναι η ψευδέστηση ότι το ενημερώνομαι και το ενημερώνει είναι κάτι πολύ απλό και αυτό το έχει δημιουργήσει το διαδίκτυο. Είναι πολύ δύσκολο να ενημερώνεται κανείς και πολύ πιο δύσκολο να ενημερώνει. Ε, εγώ συμφωνώ απόλυτα λοιπόν με τη συνάδελφο Ουάντ, η οποία έλεγε ότι πρέπει να βρούμε ένα σύστημα προκειμένου να ευνοήσουμε, να ενθαρρύνουμε και να υποστηρίξουμε πηγές αυτόνομης ενημέρωσης, ποιοτικής ενημέρωσης. Διότι σε αυτή τη μεγάλη επανάσταση των μέσων επικοινωνίας, η ανεξάρτητη ποιοτική δημοσιογραφία, η ανεξάρτητη ποιοτική ενημέρωση κινδυνεύουν να ε, ξεχαστούν από τις μεγάλες μάζες οι οποίες ανταποκρίνονται σε άλλα συμφέροντα. Επομένως, αυτή τη στιγμή το μόνο που θα μπορούσαμε να προσθέσουμε σε αυτή τη γνωμοδότηση και σε αυτή την προσέγγιση την οποία θεωρώ ιδιαίτερα σωστή είναι κάποια επισήμανση στα σημεία αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χουντής Ε, θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη γνωμοδότηση και μάλιστα παρακολουθώντας τη συζήτηση να τη συγχαρώ και να της πω να μείνει αταλάντευτη σε ορισμένες εκφράσεις που χρησιμοποιεί μέσα στη γνωμοδότηση και οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο ας πούμε κριτικής άλλων συναδέλφων και εξηγούμε στο σημείο 3 εκεί που βάζει το θέμα ότι σήμερα για τους Ευρωπαίους πολίτες είναι σημαντικό να αποκτήσουν ορθή και κριτική αντίληψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη ιστορία τη, τι αξίε και ούτω καθεξής. Και το λέω αυτό γιατί είχαμε κάνει και υπάρχει μια συζήτηση στο κατά πόσον σήμερα τα φαινόμενα που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το πώ το βλέπουν διάφοροι, αν οφείλεται ή όχι στην καλή ή ελλειπή ενημέρωση. Υπάρχει άποψη κάποιων συναδέλφων που λέει δεν υπάρχει καλή ενημέρωση στο τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιο είναι ο ρόλο των θεσμών και επομένω ε, αδίκως βλέπουμε ανθρώπους να μιλούν εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μιλούν εναντίον για τους θεσμούς ε, και επομένως υπάρχει κενό να τους ενημερώσουν. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι έτσι τα πράγματα και η έκφραση αυτή και γι' αυτό ε, την ευχαριστώ την εισηγήτρια που το βάζει αυτό ούτως ώστε να υπάρξει μια συζήτηση γιατί αγαπητοί συνάδελφοι κατά τη γνώμη μου <clears throat> η δημοκρατία θέλει πράγματι ενημερωμένους πολίτες και το πρόβλημα το ειδικό που προσπαθεί να αντιμετωπίσει η εισηγήτρια με την ε, τεχνολογία την ψηφιακή είναι ότι ενδεχομένως, μιλώ και με όρους τεχνολογικούς, αυτά τα μέσα μπορεί κάτω από ορισμένε προϋποθέσεις, με τις κυρίαρχες σήμερα προϋποθέσεις, να μην προσφέρουν ενημέρωση, αλλά να προσφέρουν πληροφορία. Αποσπασματικό, δηλαδή κάποιες γνώσεις, κάποιους αριθμούς, κάποιες δηλώσεις, που όμως δεν είναι ενημέρωση, είναι πληροφορία. Και όπως λένε οι προβληματισμένοι φιλόσοφοι, από τη στιγμή που βρήκαμε την πληροφορία χάσαμε την γνώση και την ενημέρωση. Ε, δεύτερο, διότι αυτή η αντίληψη πάει ακριβώς στο... Ο ενημερωμένος πολίτης πρέπει να είναι ενεργός. Και επομένως οι ψηφιακές αυτές πλατφόρμες ως ένα βαθμό δημιουργούν όλο και περισσότερο την ανάγκη για πιο άμεση, μορφές άμεσης δημοκρατίας. Σωστή λοιπόν, σωστός ο προβληματισμός να δούμε, όχι πάντα άμεση δημοκρατία, αλλά όχι αντιπροσωπευτική. Θα σας έλεγα όμως ότι ανασταλτικός παράγοντας αυτή την όρεξη που ανοίγει στον πολίτη είναι το γεγονός ότι ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, μετά την επικύρωση ή κατά τη διάρκεια της επικύρωσης της συνθήκης της Λισαβόνας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί εκπέμπουν αρνητικό μήνυμα για δημοψηφίσματα όσο αφορά τις, συγκεκριμένες, αυτή, ε, τις συγκεκριμένες κυρίαρχες πολιτικές και διαδικασίες που ο πολίτη ο Ευρωπαίο μιλάει για την πορεία τη Ευρώπη, για την πορεία τη χώρα και δεν μιλώ για δευτερεύοντα δημοψηφίσματα. Μια τρίτη παρατήρηση και θα τελειώσω είναι ότι εδώ πρέπει να δούμε πώς η ψηφιακή τεχνολογία, επειδή αυτό το ζήτημα συζητάμε, θα βοηθήσει όχι τη, τη δημοκρατία ως διαδικασία, τη δημοκρατία ω ουσία. Παράδειγμα, εικόνα. Το πρόβλημα που έχουμε ε, στην Ευρώπη της Δημοκρατίας δεν είναι ε, πρόβλημα δημοκρατίας, δεν είναι ότι οι διαδικασίες δεν ακολουθούνται, ότι περιστέλλονται δικαιώματα, ότι εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είμαστε εκλεγμένος θεσμός δεν μας αφήνουν πολλές φορές να αποφασίσουμε, αλλά είναι και θέματα ουσίας. Ποια, ποιας ουσίας. Ουσία είναι τι αποφασίζει καθένας μας και εν τέλει σε ποια πράγματα μπορεί να αποφασίσει ο πολίτης. Η εμπειρία η τελευταία των πρόσφατων καιρών α, επιτρέψτε μου να πω η ελληνική εμπειρία, είναι ότι όλα πια είναι αυτοματοποιημένα. Έχουν μπει σε αυτόματους πιλότους, ξεπερνάς τόσο το έλλειμμα, αυτό θα γίνεται, θα γίνεται κύρωση, δεν γίνεται καμία συζήτηση και ούτω καθεξής. Δεύτερη πλευρά. Τι αποφάσει για τέτοια κρίσιμα πράγματα για την πορεία ενό τόπου τι παίρνουν μη θεσμικά όργανα. του χάρη, περιμένουμε όλοι, εμεί και άλλε χώρε, και στο μέλλον θα περιμένουν και άλλε, τι θα αποφασίσει το Eurogroup. Τι θα πει ο κύριο Ντάιζεμπλου και τελειώνω. Εκεί δεν υπάρχει ενημέρωση. Ε, το τι συζητείτε στο Eurogroup. Περιμένουμε όλοι την καινούρια μορφή επικοινωνίας. Ένα tweet. Ε, ένα tweet, ένα Twitter, όπω θέλετε πέστε το, του κύριου Ντάζεμπλουμ να πει το κλείσαμε ή ένα tweet του κύριου Σόιμπλε ή ένα tweet του δικού μα Έλληνα Υπουργού ότι δεν το κλείσαμε και έχουμε δυσκολίε τι να ενημερωθεί ο πολίτη και τι αποφασίσαν εκεί και ποια είναι η ενημέρωση. Τι μετέπειτα, μετά γίνεται προπαγάνδα και αξιοποίηση. Επομένω, ε, εγώ νομίζω ότι ε, ε, κατά βάση συμφωνώ με τα θέματα που θίγει η συγγήτρια. Ορισμένε παρατηρήσει μπορούμε να κάνουμε, είπε και ο συνάδελφο που είμαστε από την ίδια ομάδα. Το θέμα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι πρέπει να μα απασχολήσει και επί τη ουσία για να μπορέσει η Επιτροπή μας να παίξει το ρόλο της αυτό που νομίζω είναι αναβαθμισμένος τουλάχιστον στην υπενθύμηση αρχών και αξιών που πρέπει να λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ και πάλι για την... Ευχαριστούμε πολύ. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα κάποιος να πάρει το λόγο. Να ξαναδώσω λοιπόν το λόγο στην ισχύτρια μας. Παρακαλώ, κύριε Adinolfi. Ευχαριστώ. Θα καταφέρουμε σίγουρα να εμβαθύνουμε όλα τα σημεία που επισημάνατε, τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα. Το μόνο που ήθελα ήταν να ξεχωρίσουμε τρία σημεία τα οποία εμένα απασχολούν ε, πιο πολύ σε βάθος. Πρώτα απ' όλα ένα τεχνικό ζητηματάκι. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι η αντιπροσωπευτική δημοκρατία θα αντικατασταθεί από την άμεση δημοκρατία. Εδώ έχουμε να κάνουμε το πρόβλημα της ηλεκτρονικής δημοκρατίας. Οπότε μην ξεχνάμε, μην αφαιθούμε Ας μην ξεχνάμε ότι δίπλα στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία και την άμεση δημοκρατία υπάρχουν νέα τεχνολογικά μέσα που μας δίνουν τη δυνατότητα μιας ηλεκτρονικής δημοκρατίας. Σε αυτό αναφερόμαστε σε αυτή την έκθεση. Αλλά ναι, σίγουρα και εγώ είμαι πεπισμένη ότι αντιπροσωπευτική δημοκρατία ε, υπάρχει και θα υπάρχει πάντα. σε καμία περίπτωση δεν θέλω να πω ότι θα αντικατασταθεί από την στη δημοκρατία. Απλά έχουμε τα νέα ηλεκτρονικά μέσα, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα για μεγαλύτερη συμμετοχή του πολίτη στις αποφάσεις που λαμβάνουμε στα θεσμικά όργανα. Τώρα όσον αφορά τη χειραγώγηση, και εγώ είμαι πεπισμένη ότι υπάρχουν κίνδυνοι. Γι' αυτό τον λόγο είναι σημαντικά ορισμένα πιλωτικά έργα όπως αυτό που έχει αναπτύξει το Κοινοβούλιο. Αυτά τα πιλωτικά έργα θα πρέπει να υλοποιηθούν το ταχύτερο δυνατόν ώστε να κάνουμε κάποια πειράματα. Να δούμε πώς ε, θα προσεγγίσουν τέτοια πιλωτικά έργα και οι πολίτες. Ώστε να αξισορροπήσουμε τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους και να έχουμε στη διθεσή μα ένα μέσο όσο το δυνατόν πιο αποδοτικό, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Τώρα όσον αφορά τη χειραγώγηση, φυσικά δεν την επενέσαμε εμείς, από τους Ρωμαίου αυτοκράτορες ε, μέχρι τα πλέον πρόσφατα καθεστώτα ε, Πολλοί κόσμοι κέρδισε πολλά μέσα τη χειραγώγηση των πληροφοριών. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Τώρα όσον αφορά τις σημειώσεις για τους ε, εκπαιδευτικούς και τα σχολεία και την κριτική σκέψη του πολίτη. Εγώ σε αυτή την επιτροπή τα χρόνια που δουλεύω βλέπω ότι δεν έχουμε συγκεκριμένες αρμοδιότητες παιδείας όσον αφορά τα κράτη-μέλη. Αλλά εγώ ε, πάντα θα επαναλαμβάνω σε αυτές τις επιτροπές ότι παιδεία και πολιτισμός δεν σημαίνει μόνο δεξιότητες για να μπει κανείς στην αγορά εργασίας. Γιατί, διότι στους φοιτητές, στους μαθητές της νέας γενιάς είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε μια δυνατότητα να αναπτύξουν κριτική σκέψη ώστε να έχουν τα, πολιτιστικά, τα πολιτισμικά εργαλεία και μέσα για να κάνουν ενσυνείδητες σκέψεις χωρίς να αποτελούν το αντικείμενο χειραγώγησης. Εκεί παίζουν σημαντικό ρόλο τα σχολεία, η εκπαιδευτική, όλα τα μέσα που εμείς προσφέρουμε και όλες οι πηγές που προσφέρουμε και όλα τα κονδύλια που προσφέρουμε ε, μέσω προγραμμάτων όπως το Εράσμους ε, που παρέχουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να αναπτύξουν την κριτική του σκέψη, ε, την πολιτιστική του σκέψη, όχι μόνο τεχνικές δεξιότητες. Αυτά λοιπόν. Το σύντομο δυνατόν θα στείλω, θα διαβάσω συγγνώμη τις ε, τροπολογίες που θα μου στείλετε και θα συναντηθούμε με τους και ηγητέ για τις συμβιβαστικέ τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και άλλη μια φορά. 7 Ιουνίου στις 3 είναι η προθεσμία υποβολή τροπολογιών και εδώ μπορούμε να κλείσουμε αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης και να περάσουμε στο επόμενο επενδύσει σε θέσει εργασία και ανάπτυξη, μεγιστοποίηση τη συμβολή των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Ο κ. Χουντή είναι εισηγητή για την γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και πριν του δώσω το λόγο θα ήθελα να επενθυμίσω στους συναδέλφους ότι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι 3η 7 Ιουνίου στις 11 και η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας θα λάβει χώρα στις 13 Ιουλίου. Κύριε Χουντή, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, θέλω να ευχαριστήσω τους συντονιστές και την Επιτροπή μας που μου ανέθεσαν α, αυτή τη γνωμοδότηση. Μια γενική παρατήρηση που ισχύει και για τις άλλες γνωμοδοτήσεις. διαβάζει το μισό τίτλο και είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Υπάρχει ο <laughs> υπόλοιπος τίτλος που σου βάζει τους περιορισμούς του. Αυτό είναι το θέμα θα δεις, αλλά από την άποψη πώς τα διαστρωτικά και επενδυτικά ταμεία θα συμβάλλουν σε αυτή την υπόθεση. Και εκ του γεγονότος ότι δεν κάνουμε εμείς την έκθεση, κάνουμε την γνωμοδότηση και λόγω περιορισμένου χώρου, επομένως αυτά που θα προσπαθήσω να σας πω, αυτά που έχετε δει ως ε, αρχικό σχέδιο, είναι ορισμένα σημεία που τα θεωρώ ως βάση για τη συζήτησή μας. Ε, δεν θεωρώ ότι τελειώνει αυτή η υπόθεση. Και βεβαίως δεν απηχεί το σύνολο των σκέψεων ή και των προτάσεων που έχω, ε, διότι προφανώς ε, είναι οι περιορισμοί σου δυσκολεύουν την τοποθέτηση. Έτσι ε, θεωρήστε ότι αυτή η βάση της συζήτηση στέκεται στα πιο βασικά κατά την άποψή μου θέματα που νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολήσουν στη συνέχεια της υπόθεσης, στη συνέχεια της συζήτησης, συγγνώμη, ούτως ώστε η Επιτροπή μας να καταθέσει ένα ολοκληρωμένο κείμενο, άλλωστε η γνωμοδότησή μας θα πάει στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το πρώτο που θέλω αρχικά να επισημάνω είναι ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση με την πολιτική συνοχή και τους στόχους της όπως είναι η μείωση των ανισοτήτων στις περιφέρειες και η επίτευξη μιας πραγματικής οικονομικής και κοινωνικής σύγκλησης. Ε, μια κουβέντα παραπάνω. Θυμίζω τη σημασία της πολιτικής συνοχής. Αυτό έχει αξία γιατί θα φανεί και παρακάτω. Μια πολιτική από τα καυχήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, όμως θα δούμε τους περιορισμούς ή εν πάση περιπτώσει τι μπορεί να γίνει μέσω των επενδυτικών ε, διαρθρωτικών ταμείων. Δεύτερο σημείο θα έλεγε κανείς είναι ο ρόλος που παίζουν τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία στην υλοποίηση αυτών των στόχων διότι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα ουσιαστικά αποτελούν τα κύρια μέσα για να προωθηθεί η πολιτική συνοχής και από την άλλη πλευρά ίσως και τις μοναδικές πηγές χρηματοδότησης. Τι εννοεί ο συγγραφέας ως προς αυτό, κάτι που το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ότι λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης και των πολιτικών της λιτότητας και των ακραίων κατά την άποψή μου δημοσιονομικών προσαρμογιών, οι προπολογισμοί των κρατών μελών συρρυκνώνονται. Έτσι, εθνική χρηματοδοτική πόρη για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων όλο και περιορίζονται σημαντικά. Με αποτέλεσμα οι ροές από αυτά τα ταμεία ουσιαστικά καταλήγουν να είναι ίσως και η μοναδική ροή, η μοναδική πηγή για τη χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων, ούτω ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της ε, ανάπτυξης και της απολύση των νέων και ιδιαίτερα της μείωσης των, ε, της ανεργίας. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, αφού λοιπόν τα επενδυτικά και διαρθρωτικά ταμεία, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, είναι οι μοναδικές χρηματο ε, πηγές χρηματοδότησης τέτοιων προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των θέσεων εργασία και τη ανάπτυξη και εν τέλει για την εξυπηρέτηση τη συνοχή, αφού είναι μοναδική πηγή, τότε οφείλω να σας πω, δεν περιλαμβάνεται βεβαίω, αλλά εννοείται, γι' αυτό είναι έμφαση, ότι υπάρχουν δύο περιορισμοί ως προ αυτό. Ε, τι μπορεί να περιμένει κανείς από, τα, από αυτά τα, τα κονδύλια. Τον έναν ήδη τον είπαμε και το σχολιάσαμε και σε προηγούμενη γνωμοδότηση. Ότι το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο είναι χαμηλότερο. Αυτό που τρέχει χαμηλότερο από το προηγούμενο. Επομένω υπάρχει εκεί ένα περιορισμό. Και ο δεύτερο περιορισμό, που ενδεχομένω δεν έχει μελετηθεί καλά και ίσω δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα καλά, είναι ότι τα κονδύλια, τα κονδύλια από αυτόν τον, ε, τα κονδύλια που, ε, από τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία έχουν τεθεί κάτω από την αρχή και το κριτήριο της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας μετά την ψήφιση του κανονισμού 1303, αν θυμάμαι καλά, του 2013. Επομένως, λιγότερα χρήματα από το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, μακροοικονομική αιρεσιμότητα, δηλαδή να είσαι εντάξει με δημοσιονομικούς στόχους για να μπορείς να παίρνεις αυτά τα κονδύλια. Ε, αυτό βάζει ένα φραγμό. Επομένω, αυτά που λέω και θα τελειώσω γρήγορα, ότι πρέπει να δοθεί έμφαση, είναι η μοναδική χρηματοδοτική πηγή κτλ. Ε, καταλαβαίνω ότι έχει ορισμένου περιορισμού τη συγκυρία ή τη ακολουθούμενη κυρίαρχη πολιτική. Επομένω, εδώ έχουμε αυτό το, το πρόβλημα. Ε, Τέλο, αυτό που εν πάση περιπτώσει επισημαίνει ω βάση στη συζήτησή μα, είναι κάτι το οποίο, στο οποίο συμφωνούμε, η έμφαση που πρέπει και εμεί να υπογραμμίσουμε είναι ότι έχουμε να κάνουμε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με, ένα πρόβλημα, με το πρόβλημα της νεολαίας. Σε πολλές χώρες ε, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ξεπερνάει τα πλαίσια, είναι σε πρωτοφανή επίπεδα, ίσως και πάνω από το 40% και δεν φαίνεται να αντιμετωπίζεται παρά τις κάποιες υποσχέσεις, τα κάποια προγράμματα που περιλάμβανε το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ήταν πενιχρά όπως αποδεικνύεται και η σκέψη που τίθεται στην γνωμοδότηση είναι να αξιολογηθεί αυτή, εν πάση περιπτώσει, προσπάθεια να βγουν συμπεράσματα από την πλευρά της Κομισιόν, ώστε να κατανοηθεί ότι χρειάζεται αναπροσαρμογή, θέλετε ενίσχυση, γιατί το πρόβλημα παραμένει και δεν φαίνεται να αντιμετωπίζεται με αυτά τα πενιχρά μέσα και την περιορισμένη πολιτική με την οποία ε, ή δεν είχε και κανένα αποτέλεσμα. Και το, τελευταίο, το πρώτο τελευταίο, συγγνώμη για να μην σας κουράζω, προφανώς σε τέτοια προγράμματα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Πρέπει να παίρνει υπόψη σου τις κοινωνικές αλλαγές που γίνονται μέσα στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Μιλώ για την μεταναστευτικό προσφυγικό και επομένως τα προγράμματα αυτά πρέπει να παίρνουν υπόψη ε, το θέμα της υποδοχής, υποστήριξης και ενσωμάτωσης αυτού του πληθυσμού που ενσωματώνεται στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Το τελευταίο είναι, θα έλεγε, μια υποδός η οποία αφορά και ουσία και γραφειοκρατία ότι πρέπει οι συνέργειες μεταξύ των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών προγραμμάτων και άλλων προγραμμάτων που στοχεύουν στο ίδιο σημείο να γίνουν πιο στενότερες ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικές. Αυτά και περιμένω με ενδιαφέρον προφανώς τα σχόλιά σας, τις προπολογίες σας και με τις διαδικασίες που θα εκφωνήσει το τέλος το Πρόεδρου να καταλήξουμε σε ένα συνεκτικό κείμενο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Να δώσουμε λοιπόν καταρχήν το λόγο στους κοιόδες συζητητές ε, το λόγο αν το επιθυμούν και στη συνέχεια οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Κύριος έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, άρισα λίγο γιατί πρέπει να ακούσω τη διερμηνία. Να ευχαριστήσω λοιπόν ε, τον εισηγητή για αυτήν την ε, γνωμοδότηση για την οποία ενδιαφέρομαι τόσο ο Στιώδης όσο και ο συντονιστής ε, του ΕΛΚ στο πλαίσιο της Επιτροπής για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και πάλι για το ίδιο θέμα. Ε, εμείς χαιρετίζουμε τις μεταρρυθμίσεις σε ό,τι αφορά τον ε, κανονισμό για τις κοινέ διατάξεις αφού ε, ακριβώς στοχεύουν στην καλύτερη αξιοποίηση των σχετικών ταμείων για την δημιουργία θέσεων εργασίων και την ανάπτυξη. Θα πρέπει προφανώς να γίνει μια αξιολόγηση για να δούμε και το χαιρετίζουμε αυτό να υπάρχει μια αξιολόγηση για να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα αλλά σχετική αναγίνωση έγινε πριν από πέντε μήνες πράγμα το οποίο βέβαια θέτει και κάποια ερωτήματα τελικά και δημιουργεί δυσκολίες. Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις του δικού μας στο πλαίσιο τη γνωμοδότηση. Εμεί ε, συμφωνούμε με τα όσα αναφέρει σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην ε, εκπαίδευση και στην κατάρτιση και τη διασφάλιση συνεργειών, ε, όπω ανέφερε στο τελευταίο του σχόλιο ο κ. Σιγητή, ώστε ακριβώ να αυξηθεί η αποτελεσματική αξιοποίηση των κοντιλίων των ταμείων. Ωστόσο, και γνωρίζατε ότι θα υπάρξουν και κάποια ωστόσο εδώ, εμεί σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση προγραμμάτων για την ε, ε, ε, τη χρηματοδότηση του προγράμματο για την καταπολέμηση τη ανεργία των νέων, την περισσότερη απασχόληση των νέων. Το να λέμε από τη μία πλευρά ότι θέλουμε να το υποστηρίξουμε από την άλλη, να λέμε στην ίδια παράγραφο ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα, είναι λίγο προβληματικό. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε κατά πόσο πρέπει να συνεχιστεί η χρηματοδότηση, αφόσον έχουμε προηγουμένω αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα αυτού του προγράμματος. Επίση έχουμε κάποιε συμφωνισμένε προτεραιότητε σε ό,τι αφορά αυτά τα ταμεία και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο υπάρχει η ευελιξία την οποία θα ε, θέλουμε να έχουμε για να αντιμετωπίσουμε και το μεταναστευτικό και προσφυγικό ε, πρόβλημα να σεβαστούν και τα σχετικά όρια που έχουν τεθεί και στους ε, προπολογισμού. Δεν θα πρέπει δηλαδή να συγχαίουμε και το ζήτημα ούτω ή άλλω τη προσφυγική κρίση και του προσφυγικού προβλήματο με του υψηλού αριθμού των υπολείπων μεταναστών, οικονομικών δηλαδή μεταναστών. Επίση, η Επιτροπή είπε ότι θα προβεί σε μια επανεξέταση των επιχειρησιακών προγραμμάτων για την περίοδο 2014-2020 αν υπάρξει κάποιο αίτημα από την πλευρά των κρατών μελών και αυτό είναι πολύ σημαντικό κατόπιν αιτήματο των ε, εμπλεγωμένων κρατών μελών. Οπότε δεν θα πρέπει να ξεχνάμε δηλαδή ε, πως υπάρχει ακριβώς αυτή η μακροπρόθεσμη διάσταση, αυτός ο μακροπρόθεσμος ανατολισμός ε, των ταμείων για την προώθηση της συνοχής και της ανάπτυξη Προτού δηλαδή αντιμετωπίσουμε αυτά τα κονδύλια, κάποια άλλα προβλήματα. Και επίσης οι συνάδελφοι ε, έχουν επανειλημμένα υποστηρίξει το να υπάρξει μια ε, μείωση ε, σε σχέση με το, την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Δηλαδή, εμείς δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει η Επιτροπή κάθε φορά να προτείνει μια αύξηση των σχετικών κονδυλίων. Αντιθέτως, θα πρέπει να εστιάσει στην αποτελεσματικότερη χρήση των κονδυλίων. Οπότε, αναμένουμε με ενδιαφέρον τις συζητήσεις που θα κάνουμε με την Ισχυτή και τους υπολείπους συναδέλφους, ούτως ώστε να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία μέσα στο κείμενο μεταξύ μόνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιο άλλο σκιώδη που θέλει να πάρει το λόγο. Είστε σκιώδη. Η κυρία Φερχάιν τότε καταρχήν. Ναι, θα ήθελα. Ε, Απλώ ε, ήθελα να πάρω το λόγο εκ μέρου του κυρίου Ντραγκίτση που είναι σκιώδη για το σχέδιο τη νομοδότηση. Μπορώ λοιπόν να συνεχίσω, Πρόεδρε. Καλώ. Καλησπέρα σε όλου όπως σας είπα θα παρουσιάσω α, τις απόψεις ε, του κύριου Ντραγκίτση ό,τι αφορά το σχέδιο γνωμοδότησης, ο οποίος ε, βλέπετε πως απουσιάζει. Ε, όπως έδειξε η έρευνα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, ε, βλέπουμε να σημειώνεται μία ήπια οικονομική ανάπτυξη το 2015, αλλά τα κοινωνικά ζητήματα και η ε, εφαρμογή των σχετικών μεταρρυθμίσεων βρίσκονται σε πολύ διαφορετικά επίπεδα ανά κράτος μέλος. Οπότε θα ήθελα εδώ να επισημάνω κάποια επιχειρήματα του κ. Ντραγκίτσε Υπάρχουν λοιπόν διαφορέ ανάμεσα στα κράτη-μέλη παρά τι προσπάθειε που έχουν γίνει και κάποιε από αυτέ τι διαφορέ αυξάνονται. Επίση, η μακροπρόθεσμη ανεργία, ειδικότερη ανεργία μεταξύ των νέων, παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Και ε, τα όσα γίνονται σε επίπεδο μέτρων για την εκπαίδευση δεν επαρκούν. Και ε, κάτι ακόμα, η ε, τρέχουσα μεταναστευτική κρίση δημιουργεί και κινδύνου σε ό,τι αφορά τι και δημιουργεί και περαιτέρω ε, προκλήσει ε, για τι ε, κοινωνίε μα και τα συστήματα παιδεία μα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ενισχύσουμε με κάθε δυνατό τρόπο τη συνοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά συνέπεια η περιφερειακή κοινωνική συνοχή θα πρέπει να βρεθεί στον πυρήνα τη Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 έτσι ώστε όλα, όλοι οι πόροι που έχουμε στη διάθεσή μα να αξιοποιηθούν για την εφαρμογή αυτή τη στρατηγική. Ε, τα ε, διαφθορτικά και επενδυτικά ταμεία αποτελούν τον κύριο ε, μέσο για την εφαρμογή τη πολιτική συνοχή και επίση αποτελούν σημαντικό τμήμα του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη και συμπληρώνω το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Από το 2014 ε, ε, υπάρχει ένα μεταρρυθμισμένο πλαίσιο ε, για τα επενδυτικά και διαρθρωτικά ταμεία με απλουστευμένες κανονές, απλουστευμένες διαδικασίες, περισσότερο εστιασμό στα αποτελέσματα και πιο στοχευμένα θεματικά πεδία. Παρόλα αυτά, παρόλε αυτέ τι μεταρρυθμίσεις, καποια κάποια κράτη-μέλη δεν είναι σε θέση να αξιοποιήσουν πλήρω αυτέ τι νέε δυνατότητε και χρειάζονται περισσότερη καθοδήγηση. Η ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο καθώς αποτελεί το κυριότερο διαθωτικό ταμείο που αγγίζει άμεσα τις ζωές ε, των πολιτών. Ε, δηλαδή αφορά τόσο εργαζόμενους, ανέργους, άτομα που, έχουν, που δεν συμμετέχουν εργά στην κοινωνία, ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, όλοι αυτοί λοιπόν εποφελούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και κατά συνέπεια το Ταμείο αυτό θα πρέπει να αξιοποιηθεί στο μεγαλύτερο ε, ε, δυνατό βαθμό ε, για προγράμματα τα οποία υποστηρίζουν και το τομέα της εκπαίδευσης και ειδικότερα των εκπαιδευτών. Αυτό στο μέσα θα πρέπει να υποστηριχθεί και στο πλαίσιο των πορισμάτων της, της έκθεσης παρακολούθησης για το τομέα της παιδείας προσθέσεως του 2015 που και που αναφέρεται ότι το να η, η, σχέση με τα επιθυμητά αποτελέσματα των, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ε, βελτιωθεί περαιτέρω. Επίσης, ε, ε, ε, μέσα στο 2016 σε ό,τι αφορά την οικονομική ανάπτυξη και τη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω τη ε, παιδεία ε, καταδεικνύει ακριβώ ότι θα πρέπει, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για επενδύσει στην εκπαίδευση και στην ε, επαγγελματική κατάρτιση, ούτω ώστε να επιτύχουμε μια εύρυθμα λειτουργούσα αγορά εργασία. Όπω αναφέρει και ο ίδιο ο εισηγητή, οι οικονομικοί και κοινωνικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από, την, ακριβώς, ε, από τις ελλειπείς επενδύσεις των 100 μελών στην παιδεία παραμένουν, οπότε θα πρέπει να ε, περάσουμε ενισχυμένα το μήνυμα ότι η παιδεία αποτελεί ε, το καλύτερο, το, το πιο σημαντικό τρόπο για την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, οπότε θα πρέπει να αξιοποιήσουμε με καλύτερο δυνατό τρόπο τις δυνατότητες που μας δίνουν τα διαφθορτικά και επενδυτικά ταμεία σε συνεργασία και με άλλα προγράμματα και άλλα χρηματοδοτικά μέσα, όπω για παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατηγικών ε, Επενδύσεων και το Erasmus Plus. Επίση, ο κύριο Δραγίτση θα ήθελε να ε, τονίσει ότι ε, παρότι το τμήμα της κουλτούρας δεν αντιμετωπίζεται ως ζήτημα θεματικής προτεραιότητας μέσα στο στρατηγικό πλαίσιο του 2020, ε, αναγνωρίζεται όλο ένα και περισσότερο ο πολυδιάστατος ε, χαρακτήρας ε, του πολιτισμού και υπάρχει μια πολύ σημαντική ανάγκη να σχετίσουμε τον πολιτισμό με την, και με τον τομέα του τουρισμού και να αξιοποιήσουμε καλύτερα αυτόν τον τομέα, ούτως ώστε να συμβάλλει στην δημιουργία της κοινωνίας γνώσης και να αυξήσει την ε, συνοχή αλλά και να υποστηρίξει τις ε, ε, κεντρικές και περιφερειακές αρχές στα κράτη-μέλη, ώστε να ε, συμπεριλάβουν τα σχετικά θεματικά παιδεία στι αναπτυξιακέ του στρατηγικέ. Ε, Τέλο, ο κύριο Δραγκίτση συμφωνεί με τον εισηγητή ότι ε, το, το ζήτημα των μεταναστών και προσφύγων και των ετούντων άσυλο και επιπτώσει σε ό,τι αφορά και την αγορά εργασία δημιουργεί μία σειρά από προκλήσει και κατά συνέπεια χρειάζεται να, να υπάρξει και κατάλληλη χρηματοδοτική υποστήριξη. Ε, πέραν ε, ε, τη υποστήριξη από τα επενδυτικά και διαφορετικά ταμεία και ειδικότερα το Ταμείο Συνοχή, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αξιοποιήσουν περαιτέρω προγράμματα και περισσότερο ταμεία, ειδικότερα το Ταμείο για την υποστήριξη των πλέον ευάλωτων ομάδων, όπω και το Ταμείο για το Άσυλο ε, και την ε, ένταξη. Ο κ. Δαγκίτση θεωρεί ότι ε, μπορεί να διατυπωθεί ακόμα καλύτερα το σχέδιο νομοδότησης, οπότε αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την μελλοντική συνεργασία για την βελτίωση του σχεδίου γνωμοδότηση με τον κύριο Χουντή και του υπόλοιπου αισιώδε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η πρόεδρο, η κυρία Σφεχάιν. έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σχολιάσω δύο στοιχεία εδώ, διότι να. Ε, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ε, όταν λέμε ότι διασφαλίζοντας περισσότερα κοντήλια μπορούμε να καταφέρουμε περισσότερα. Θα πρέπει να, τα εν λόγω κοντήλια να αξιοποιούνται αποτελεσματικότερα. Οπότε εμεί θέλουμε να θέσουμε περισσότερο έμφαση στην ποιότητα των ε, ε, προκηρύξεων γενικότερα των ε, ε, δημοσίων συμβάσεων να δούμε ποιε είναι οι διαδικασίε που ακολουθήθηκαν μέχρι τώρα, υπήρξαν αποτελεσματικέ και ποια είναι τα project τα οποία χρηματοδοτούνται. Έχουν πραγματικά τα προηγούμενα project οδηγήσει στην δημιουργία θέσεων εργασία. Μήπω, για παράδειγμα, οι προκηρύξει για υποβολή προσφορών θα πρέπει να αλλάξουν σε ό,τι αφορά το περιεχόμενό του ακριβώ για να επιτύχουμε περισσότερα αποτελέσματα. Αντί λοιπόν να λέμε μόνο χρειαζόμαστε περισσότερα κονδύλια, θα πρέπει να δούμε ποιοτικά κάτι μπορεί να γίνει για να βελτιώσουμε τα πράγματα. Να δούμε δηλαδή ε, αυτά τα προγράμματα είναι προσβάσιμα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί αυτέ μεταξύ άλλων θα είναι οι μικρομεσαίε επιχειρήσει ε, οι οποίε θα κληθούν να δημιουργήσουν θέσει εργασία. Και τι έγινε με προηγούμενα τέτοια project, δημιούργησαν πράγματι θέσει εργασία. Πώ ακολουθήθηκαν αυτέ οι διαδικασίε, τι γίνεται σε σχέση με ορισμένε περιφέρειες Εάν δηλαδή δεν έχει ε, διαρθρωθεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα αναπτυξιακό για μια περιοχή, δεν μπορεί να βοηθήσει και σε τίποτα το να ε, δίνουμε απλά περισσότερα κονδύλια, να διαθέτουμε περισσότερα κονδύλια. Επίση, θα πρέπει να δούμε πιο συγκεκριμένα κατά πόσο ο πολιτισμικό και δημιουργικό ε, τομέα, ο οποίο αποτελεί και κυριτήρια δύναμη για την οικονομία, λαμβάνεται υπόψη στα εν λόγω προγράμματα. Και βέβαια ο λόγο στο μέσα αποτελεί και δική μα αρμοδιότητα και γι' αυτό ενδεχομένω θα πρέπει να τονίσουμε ακριβώ αυτό το γεγονό ότι δηλαδή θα πρέπει να συμπεριληφθεί ο τομέα του πολιτισμού και τη ε, ε, δημιουργία ε, σε τέτοιου είδου προγράμματα για τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασία. Και το ζήτημα των επενδύσεων στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση αφορά βέβαια και ένα ζήτημα του πώ ε, συντονίζουμε μεταξύ του διαφορετικά προγράμματα. Εάν δεν είναι σωστά συντονισμένα μεταξύ του ε, τα προγράμματα, ε, μπορούμε αντί να διορθώσουμε κάποια προβλήματα, ακριβώ να τα οξύνουμε ακόμα περισσότερο. Οπότε, οπότε θα πρέπει όταν λέμε πώ ακριβώ μπορούμε καλύτερα να συνδέσουμε αυτά τα κονδύλια και πώ αξιοποιούμε αυτά καλύτερα αντί να λέμε μόνο και πάντοτε ότι θέλουμε απλά περισσότερα κονδύλια και περισσότερη χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, ο e, Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω με ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Η έκθεση αναφέρει πολύ σημαντικά ζητήματα, αλλά έχω ένα πρόβλημα με την αιτιολόγηση για αυτή την επιτροπή που θα έχει πόρους από διάφορες πηγές. Το Ευρωπαϊκά Δραστηριοτικά Ταμεία ε, με τη βοήθεια περιφερειακών ταμεία είναι διαφορετικές ε, ταμεία χρηματοδότησης που έχουν τελείως διαφορετικούς στόχους και τρόπους χρηματοδότησης και η δήλωση ότι η πολιτική συνοχή είναι η μόνη πηγή χρηματοδότησης αυτών των προγραμμάτων δεν είναι σωστή. Δεν είναι η μόνη πηγή, είναι ίσως η πιο σημαντική, αλλά όχι η μόνη. Επίσης, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι η πολιτική συνοχής ε, έχει τις εθνικές κυβερνήσεις να έχουν τις πιο, τον πιο σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, η εθνική πρικοδότηση ε, καθορίζεται ε, βάσει της ε, χρήσης των κονδυλίων ε, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για συγκεκριμένους σκοπούς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποδιαιρεί σε πακέτα τα κονδύλια, αλλά το περιεχόμενο των πακέτων σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τα ε, χώρες μέλη. Και υπάρχουν τα εξή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρχάς δεν πρέπει να δεχτεί όλες τις προσδοκίες που υπάρχουν στο πακέτο της διαπραγμάτευσης. Δεν υπάρχει όμως το αντίθετο. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να συμπεριλάβει κάτι στον εθνικό κορβανά το οποίο δεν επιθυμεί μια κυβέρνηση. Όταν αναφερόμαστε σε πολιτική συνοχή, θα πρέπει να ε, δούμε και την κατάσταση της κρίτησης. Αυτή τη στιγμή βιώνουμε μια πολύ παράδοξη και ιδιαίτερη κατάσταση. Υπάρχουν κυβερνήσεις οι οποίες για χρόνια, ε, παρά τις διάφορες προεκτικές, δεν υπέβαλαν ποτέ προγράμματα τα οποία ε, προορίζονταν για όσα προβλέπονται σε αυτή τη γνωμοδότηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να δημιουργήσουμε προσδοκίες οι οποίες θα αποτελέσουν στη συνέχεια έναν ελάχιστο κοινό παρονομαστή και θα δώσουν τη δυνατότητα στα προγράμματα τα οποία αναφέρονται στη γνωμοδότηση να υλοποιηθούν. Εάν αυτή τη στιγμή ο πολιτισμός, ε, η παιδεία ε, και το ορίζοντας 2020 σε μεγάλο βαθμό καλυφθούν και από το πρόγραμμα Juncker και επομένως καλύψουμε τις απαιτήσεις για την επαιδεία και τον πολιτισμό, θα πρέπει να μην λησμονούμε ότι πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες συνέπειες όσον αφορά, για παράδειγμα, την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν επενδύσεις, ε, όπω είπε και η συνάδελφο, που να γίνονται προ αυτή την κατεύθυνση. Αλλά επίση δεν υπάρχει και κατάλληλη αξιολόγηση για το κατά πόσον γίνεται αποτελεσματική χρήση ε, και αν πραγματικά είναι εφαρμοσμένο και προσαρμοσμένο στην αγορά εργασίας. Ε, αυτή τη στιγμή ε, δίνονται 10 δις ευρώ σε διάφορα προγράμματα και σε κάποιες περιπτώσεις 10 εκατομμύρια ευρώ οδήγησαν στην απασχόληση χιλίων ατόμων. Σε ορισμένε φορέ μόνο 5-10 άτομα απέκτησαν μια θέση εργασία με αντίστοιχη ε, επένδυση. Επομένως, στην περίπτωση των μεγάλων επενδύσεων, σε κάθε συμφωνία περιγράφονται κάποιες ε, ε, προϋποθέσεις όσον αφορά την αύξηση της απασχόλησης κατά ένα συγκεκριμένο ποσοστό ατόμων. Πρέπει λοιπόν να αξιολογήσουμε κατά πόσον αυτές οι προσδοκίες οι οποίες υποδεικνύονται στις Γενικές Συμφωνίες γίνονται σεβαστές στη συνέχεια. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε τη διαπραγμάτευση της τύπητη, που δεν είναι βέβαια αρμοδιότητα της Επιτροπής μας. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα άνοιγμα των ε, ε σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ και ξέρουμε ότι αν υπάρξει συμφωνία, κάποιοι τομείς θα υποφαληθούν ενώ κάποιοι άλλοι θα πληγούν. Ο πολιτισμός εξαιρείται από αυτή τη συμφωνία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρχουν, δεν θα υπάρχουν συνέπειε έμεσε, είτε θετικές είτε αρνητικές από αυτή τη συμφωνία. Επομένως, θα πρέπει να επισημάνουμε ίσως ότι ο πολιτισμός θα πρέπει να προστατευτεί μέσω της πρόσβασης σε μέσα ή σε επενδύσεις ε, χάρη στις οποίες οι πιο ευαίσθητοι τομείς, όπως είναι η παιδεία και ο πολιτισμός, δεν θα υποστούν αρνητικές συνέπειες ε, από αυτή την, το άνοιγμα και σε υπηρεσίες ε, γιατί αν έχουμε άνοιγμα υπηρεσιών από τις Ηνωμένε Πολιτείες προς την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υπάρχει απειλή για την παιδεία αλλά και για όλα τα καλλιτεχνικά ε, στοιχεία στην Ευρώπη. Εμείς θέλουμε να συνεχίσει αυτή η υποκυλομορφία, ο πολιτιστικός πλούτος και ξέρουμε ότι το Ταμείο αυτό θα μπορούσε ίσως ε, να προστατεύσει όλα όσα θα μπορούσαν να εξαφανιστούν ή να υποστούν πιέσεις οι οποίες δεν θα είναι προς όφελος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατόπιν. Αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε τις κατηγορίες που προτείνεται, να υπενθυμίσω στον ε, εισηγητή ότι η πολιτική συνοχή είναι πολύ δημοφιλής και αυτό γιατί πολύ συχνά οι κυβερνήσεις ζητούν υποστήριξη για προγράμματα τα οποία ε, δίνουν υποστήριξη σε κυβερνητικό επίπεδο και σπανίως υποστηρίζουν προγράμματα σε επίπεδο τοπικών και περιφερειακών αρχών. Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο ίσως θα έπρεπε να τονίσουμε στη γνωμοδότηση. Το γεγονός ότι τα πιο αποτελεσματικά ε, κονδύλια, αυτά τα οποία δαπανώνται, είναι όσο χαμηλότερο είναι το επίπεδο και όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο ελέγχου αυτών των δαπανών. Ευχαριστώ κυρία Τρούπη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ στο τελευταίο ζήτημα αυτά που έχουμε εμείς αποφασίσει ως προϋποθέσεις, δηλαδή σε ό,τι αφορά τις εξαιρέσεις, σε ό,τι αφορά τα οπτικοακουστικά ε, μέσα και τον ε, κλάδο του πολιτισμού, ο εν λόγω κίνδυνο ο οποίο αναφέρθηκε μόλι τώρα δεν υπάρχει. Οπότε θα πρέπει εμεί πραγματικά να επιμείνουμε σε αυτό. Δηλαδή στο να διαπραγματευτεί η Επιτροπή με βάση την εντολή που τη δώσαμε και του περιορισμού που θέσαμε. Άρα λοιπόν από αυτό θα εξαρτηθεί το, το κατά πόσο υπάρχει ένας κίνδυνος ε, εδώ γιατί ακριβώς εμείς εγκαίρως είχαμε τονίσει της δικές μας επιφυλάξεις ε, και προβήκαμε. Ε, στι κατάλληλε ουσιασίε ε, στην Επιτροπή. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα εδώ, να πω ότι είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα διαστοτικά και επενδυτικά ταμεία θα πρέπει να καταστούν πιο γνωστά και στα ίδια τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει είναι και εξακολουθεί να συμβαίνει ότι μεταξύ των διαφορετικών αναπτυξιακών προγραμμάτων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει διαφορετικό επίπεδο γνώσης τους από την πλευρά των διαφόρων διούχων. Οπότε ε, και αυτό που αναφέρεται εδώ είναι πολύ σημαντικό ότι δηλαδή ο συντονισμός, οι συνέργειες μεταξύ αυτών των διαφορετικών προγραμμάτων ε, και των ταμείων με άλλα ταμεία δεν είναι τόσο ανεπτυγμένο όσο θα έπρεπε. Και οι διάφορε συμβουλευτικέ υπηρεσίε, δηλαδή οι αρμόδιε αρχέ των κρατών μελών, θα πρέπει και αυτέ να ορίζουν κατά πόσο υπάρχουν άλλα προγράμματα και ποια είναι, ώστε να διασφαλίζονται ακριβώς αυτές οι συνέργειες ήδη κατά τη φάση της υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ. Um, thank you very much. Στον εκπρόσωπο, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Δεν έχω να προσθέσω πολλά στη συζήτηση. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για μας. Θα ήθελα να αναφερθώ στο τελευταίο σημείο στην ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των διαφόρων ταμείων. Αυτό προσπαθούμε σε αυτή την προγραμματική περίοδο και στην επόμενη. Είναι σημαντικό επίσης να ενισχύσουμε και την αίσθηση οικειοποίησης των τοπικών αρχών και των περιφερειακών αρχών όσον αφορά ε, τα ευρωπαϊκά κονδυλία για σχετικές δραστηριότητες. Να σημειώσω επίσης ότι η πρωτοβουλία για το κλίμα έχει διάφορες δραστηριότητες παρότι φυσικά ε, λόγω των συνθήκων σήμερα στην Ευρώπη είναι δύσκολο να δημιουργηθούν ε, θέσεις εργασίας αλλά αυτή η πρωτοβουλία πραγματικά βοηθά πολύ κόσμο να ξαναβρει μια θέση εργασίας να ξαναμπεί στην αγορά εργασίας ή να βρει την πρώτη δουλειά και αυτό αποτελεί ε, και, σχετίζεται και με τις πολιτιστικές δραστηριότητες. Και έτσι χρησιμοποιούνται τα κονδύλια για τις πολιτισμικές δραστηριότητες και πολιτικές δραστηριότητες φυσικά βάσει και των ε, πολιτικών επιλογών των κρατών μελών. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω ξανά το λόγο στον εισηγητή μα, τον κύριο Χουντή, παρακαλώ. Ε, Σα ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ όλου του συναδέλφου και τι συναδέλφισε που πήραν το λόγο ε, και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις ήταν ε, πολύ καλά προετοιμασμένοι, πράγμα που είναι κολακευτικό για ένα κείμενο που έδωσε ως βάση για συζήτηση. Και επομένως ε, ε, υπάρχει περιθώριο γραπτά πια με τις τροπολογίες να δούμε πού μπορούμε να συγκροτήσουμε ένα περιεκτικό κείμενο. Απλώς θα ήθελα ε, πράγματι να προσεγγίσουμε ορισμένα θέματα που εθίγησαν ε, ως θέματα αρχής. Ε, από τις συζητήσεις βλέπω ότι έχουμε δύο διλήμματα. διλήμματα. Το ένα είναι περισσότερα χρήματα γιατί είναι λίγα όπως παρουσιάζει η εισήγηση υπάρχουν περιορισμοί ή καλύτερη αξιοποίηση των υφισταμένων. Φαντάζομαι η απάντηση για όλους μας είναι και τα δύο. Και τα δύο. Όμως δεν μπορούμε μετά από ένα όριο να μιλάμε μόνο για την αξιοποίηση των υφισταμένων κονδυλίων. Διότι κατά την άποψή μου είναι έτσι κι αλλιώς περιορισμένες οι δυνατότητες. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα το λύσουμε. Θα το δούμε προς τα που πάει αυτό το πράγμα. Και το δεύτερο ε, δίλημα που εμφανίζεται είναι πώς κρίνουμε την αποτελεσματικότητα κάποιων προγραμμάτων και τα αποτελέσματα. Ε, Παραδείγματο χάρη, στην περίπτωση που λέμε ότι πρέπει αυτά τα προγράμματα και ιδιαίτερα σε ευαίσθητου τομεί, αυτό πρέπει να τονίζεται ομολογώ περισσότερο εκπαίδευση, πολιτισμό, να δημιουργούν θέσει εργασία ε, και το ερώτημα, επειδή ετέθηκε και από την άποψη τη ποιότητα, τι εννοούμε νέε θέσει εργασία. Εννοούμε πλήρου απασχόληση με πλήρη, ας το πούμε, ασφαλιστικά δικαιώματα ή αυτές τις θέσει θέσεις που αριθμητικά σου δίνουν ε, την αίσθηση ότι έχεις κάποιο αποτέλεσμα, αλλά δεν είναι το αποτέλεσμα αυτό. Άλλωστε και τα στοιχεία λένε ότι έχουμε μια μακροχρόνια ε, ανεργία των νέων. Τέλος, δεν θέλω να πω... Ε, ναι, ένα σχόλιο λίγο για το TTIP. Θυμάμαι ή στην προηγούμενη ή σε μια πιο προηγούμενη συνεδρία της Επιτροπής μας είχε τεθεί ένα θέμα να εκπονηθεί, αν θυμάμαι καλά διορθώστε με, ε, μια έκθεση αν και ποια είναι η επίδραση, τι έχει συμφωνηθεί επ' περιπτώσει στα πλαίσια της Διατραντικής Συμφωνίας στον τομέα που μας αφορά εδώ στην Επιτροπή. Ε, και τότε είχε αποσαφινιστεί ότι έχουν εξαιρεθεί οπτικοακουστικά και άλλα μέσα και εγώ νομίζω ότι εδώ τώρα έχουμε ένα πρόβλημα ποιος είναι ενημερωμένος, τι ακριβώς συζητείται από αυτού του θέματος. Ελπίζω και με τις προτάσεις που έχουν γίνει και με τις, τα κινήματα που έχουν διαμορφωθεί ιδιαίτερα τα κινήματα στον χώρο του πολιτισμού έναντι των συνεπειών ε, δυσμενών συνεπειών για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό έτσι φαίνονται τα πράγματα να αποτρέψει να έχουμε στη γνωμοδότηση άλλωστε στη γνωμοδότηση τι μπορεί να πει σε αυτό είναι η γενικότερη προσπάθεια που κάνουμε ούτω ώστε ε, κατά τη γνώμη μου ότι TIP πρέπει να μάθουμε τι γίνεται και πάση περιπτώσει να επισημάνουμε και να χτυπήσουμε το καμπανάκι το τι θα υφίσταται ο ευρωπαϊκός πολιτισμός με την ευρύτερη έννοια μέσα από αυτή τη συμφωνία. Ε, και πάλι ευχαριστώ πολύ. Ε, περιμένω τις γραπτές προτάσεις ή και τις συνεργασίες τους, ώστε από ό,τι φαίνεται ένα κείμενο ή μια γνωμοδότηση που έχει ενδιαφέρον να την κάνουμε όσο γίνεται καλύτερη και να εκφράζει την Επιτροπή μας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Χουντή για αυτά τα πολύ ακριβή συμπεράσματα και για την εξαιρετική συζήτηση. 7 Ιουνίου στις 11 το πρωί είναι η προθεσμία υποβολή τροπολογιών. Μπορούμε λοιπόν να κλείσουμε αυτό το σημείο της ημερησίας διάταξης και φτάνουμε στο τελευταίο σημείο της σημερινή συνεδρίαση στην προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσει προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Η συγγήτρια είναι η κυρία Κάμερα Εβέρτ που συντάσσει τη γνωμοδότηση για την Επιτροπή μας. Χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες θα ήθελα να παρουσιάσω εν συντομία αυτή τη γνωμοδότηση, η οποία ουσιαστικά σχετίζεται με μια άλλη σημαντική οδηγία που παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα από την Επιτροπή την οδηγία για τα οπτικοακουστικά μέσα και τις σχετικές υπηρεσίες. Οι δύο αυτοί φάκελοι σχετίζονται στενά. Για στρατηγικούς λοιπόν λόγους, ο εισηγητής θέλει να εγκριθεί η γνωμοδότηση των συντομότερων δυνατών. Γι' αυτό προτείναμε ως προθεσμία υποβολής τροπολογιών την Τετάρτη 1η Ιουνίου στις 12 η ώρα. Διάφοροι όμως συναδέλφοι διαφωνούν με μια τόσο σύντομη προθεσμία. Θα ήθελα να μιλήσουν οι συναδέλφοι από αυτού όταν θα λάβουν το λόγο. Και δίνω τώρα το λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Κάμερεβερτ. Ja, vielen herzlichen Dank. Σας ευχαριστώ, θερμά Πρόεδρε. Θα αναφερθώ στο ζήτημα της ε, προθεσμίας ε, στο τέλος της ε, παρουσίασής μου. Καταρχήν θα ήθελα λοιπόν να εστιάσω στο περιεχόμενο αυτής της πράξεις για την προσβασιμότητα του Accessibility Act που βέβαια ε, στοχεύει στην εφαρμογή ε, των όσων προβλέπει η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με την αναπηρία και την προσβασιμότητα. Ε, στο πλαίσιο λοιπόν εδώ αυτή τη πρόταση καλύπτονται όλα τα οπτικοακουστικά μέσα συμπεριλαμβάνων και των ηλεκτρονικών βιβλίων. Οπότε εγώ εδώ κάλυψα στη δική μου γνωμοδότηση όλα αυτά κομμάτια. Δηλαδή έχουν διαγραφεί από το συγκεκριμένο σημείο και οι αναφορές αναφορούν οπτικοακουστικά μέσα και ηλεκτρονικά βιβλία. Αυτό λοιπόν που προτείνω εγώ είναι να υπάρξει μια εξαίρεση ε, σε ό,τι αφορά τους κανόνες αυτής της οδηγίας για αυτά τα δύο ε, κομμάτια. Αλλά σε ό,τι αφορά ε, τις συσκευές ανάγνωσης, ή συσκευές λήψης, αυτές δεν νομίζω πως θα πρέπει να ε, τις πειράξουμε καθόλου γιατί νομίζω πως θα πρέπει να κάνουμε εδώ μια διάκριση, αυτή διάκριση ανάμεσα στο περιεχόμενο αφενός και ανάμεσα στα μέσα πρόσβαση σε αυτό το περιεχόμενο. Αν θέλετε. Οπότε, ε, σε ό,τι αφορά τις συσκευές λήψης δεν έχω προτείνει κάποιες τροποποίησεις στην πρόταση οδηγίας της Επιτροπής. Οι δικέ μου λοιπόν προτάσει με πιο σκεπτικό γίνονται. Ακολουθούμε πολύ συστηματική προσέγγιση εδώ και είμαι βαθύτατα πεπισμένο ότι θα επιτύχουμε αποτελεσματικότερε αλλά και πιο ευέλικτε ε, λύσει ε, εάν προβούμε στι αντίστοιχε εντροποποιήσει ε, σχετικέ οδηγίε. Σε ό,τι αφορά τι υπηρεσίε οπτικοακουστικών μέσων, θα πρέπει να υπάρχουν οριστικές διατάξεις, την ίδια δηλαδή αυτή την οδηγία AVMS, και ήδη υπάρχουν, ε, έχει υποβληθεί μια πρόταση ε, για την αναθεώρησή της, της σχετικής οδηγίας, οπότε νομίζω πως αποτελεί μια ε, καλή ευκαιρία εδώ το να, έχουμε, να περάσουμε πιο κατηγορηματικά μηνύματα, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το κανονιστικό πλαίσιο για την προσβατισμότητα των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Το ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να προστατεύσουμε την ελευθερία του τύπου, τον πλουραλισμό και τα συναφή ζητήματα νομίζω πως θα πρέπει να καταστούν συνεκτικά και με το ζήτημα της προσβασιμότητας και ακριβώς ε, αυτό το ζήτημα μπορούμε να το ρυθμίσουμε με τον κατάλληλο τρόπο στο πλαίσιο αυτής της οδηγίας. Ε, ιδιαίτερα ε, σημαντικό σε αυτό το πλαίσιο είναι το άρθρο 7 της οδηγίας που καλεί τα κράτη-μέλη να αξιώνουν ε, τις υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά τους παρόγους αυτών των υπηρεσιών και των συσκευαστές των σχετικών προϊόντων σε ό,τι αφορά τη λήψη υπόψη ατόμων με αναπηρία. Νομίζω πως είναι πολύ γενικόλογη αυτή η αναφορά, δηλαδή θα πρέπει να έχουμε ε, κριτήρια προσβασιμότητας με συγκεκριμένα benchmarks και να υπάρχει και σύστημα παρακολούθηση επιτήρησης, δηλαδή σε επίπεδο κρατών ε, μελών. Κάτι τέτοιο θα πρέπει να εφαρμοστεί στο πλαίσιο της οδηγίας αυτής για τα οπτικοακουστικά μέσα και θα αποτελούσε μια ε, βελτίωση σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τα όσα ε, προβλέπονται στο, στην πρόταση οδηγίας που έχουμε μπροστά μας η οποία είναι πολύ περιοριστική από την πλευρά της. Ε, θα πρέπει δηλαδή με, με αυτές τις προτάσεις που κάνουμε θα, θα καταφέρουμε να έχουμε ακριβώς την απαραίτητη ευελιξία για, την, για τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα σχετικά άτομα στα οποία αφορά. Θα πρέπει δηλαδή να εστιάσουμε σε αυτά τα ζητήματα στο πλαίσιο αυτής της πολύ εξειδικευμένης οδηγίας για οπτικοακουστικά μέσα και όχι στο πλαίσιο μιας γενικότερας ε, ε, οδηγίας. Επίσης να θυμώσουμε ότι έχει ε, υπογραφεί από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο η σύμβαση για τα άτομα με αναπηρία αλλά και η σύμβαση σε ό,τι αφορά τον πλουραλισμό ε, των ε, μέσων ενημέρωσης. Οπότε ε, θα πρέπει εδώ να υπάρξει μια ισορροπία. Για παράδειγμα, η προσβασιμότητα σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρονικά βιβλία μπορεί να διασφαλιστεί από την πλευρά των ίδιων των κρατών μελών χωρίς να υπάρξει καμία, χωρίς να υπάρχει καμία ανάγκη να δραστηριοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε πραγματικά εδώ νομίζω πως πρόκειται για μια περίπτωση όπου θα πρέπει να σεβαστούμε την αρχή της επικουρικότητας. Δεν θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης ε, κάτι ακόμα. Σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας εφαρμογής των ε, σχετικών διατάξεων από την πλευρά των επιχειρήσεων, ε, συντάσσοντας κάποιο μια ε, επιστολή όπου ζητάει συγγνώμη μπορεί ουσιαστικά να αποφύγει οποιασδήποτε επιπτώσει, γιατί η ίδια οδηγία δεν αναφέρει κανένα είδου κυρώσει. Ε, τι προβλέπετε δηλαδή σε περίπτωση που κάποιος δεν τηρήσει τις σχετικές ε, προϋποθέσεις προσβασιμότητας, ποιος θα είναι εκείνος ο οποίος θα προβαίνει στον έλεγχο που, θα, που ακριβώς θα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ε, κάποιο προϊόν ή υπηρεσία, ποιος θα είναι ο αρμόδιος για να προβαίνει σε αυτή την αξιολόγηση, ποιος θα είναι εκείνος ο οποίος θα επιτηρεί ε, την ε, συμμόρφωση με αυτή την προσβασιμότητα, όλα αυτά δεν αναφέρονται εδώ. Γίνονται προσπάθειες τυποποίησης των τερματικών συσκευών, για παράδειγμα ηλεκτρονικά ε, ηλεκτρονικές συσκευές ε, ανάγνωση, τηλεοράσει και ό,τι καθεξής, αυτά πράγματα πράγματι ακούγονται πολύ λογικά. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι τέτοιου είδους ε, περιοριστικοί κανόνες ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων και των ηλεκτρονικών βιβλίων, ε, μπορεί να σημάνει ότι δεν θα υπάρξει παραγωγή των σχετικών ε, προϊόντων και υπηρεσιών εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν δηλαδή ε, κανεί παράγει μία ταινία και θα πρέπει στη συνέχεια να λάβει υπόψη και ευρωπαϊκού τύπου διατάξει. και διατάξεις από την πλευρά μέλους για παράδειγμα ε, και θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, προβλέψει και τους σχετικούς υποτυπωποιημένους υπότιτλους ή οτιδήποτε άλλο ε, τι θα σημαίνει ότι θα είναι τόσο ακριβή η παραγωγή μιας τέτοιας ταινίας ούτως ώστε να μην να μετατεθεί αλλού η παραγωγή, δηλαδή να επιλέγουν οι παραγωγοί να μην προβαίνουν στην παραγωγή τέτοιων ε, προϊόντων εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα επικρεμάται πάντοτε δηλαδή να δαμόκλειο σπάθη ακριβώ των διαφορετικών διατάξεων που θα πρέπει να εφαρμόσουν. Προφανώ δηλαδή είναι σωστή η, η προσέγγιση, η πρόθεση εδώ ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε την προσβασιμότητα σε ό,τι αφορά οπτικοακουστικά μέσα, αλλά ο δρόμο που ακολουθεί ε, η Επιτροπή σε σχέση με αυτό το ζήτημα είναι εσφαλμένο, οπότε θα πρέπει να δούμε πώ μπορούμε να ρυθμίσουμε αυτά τα ζητήματα στο πλαίσιο τη οδηγία ε, για τα οπτικοακουστικά μέσα, αντί να ακολουθούμε μια τόσο γενικόλογη προσέγγιση. Ε, σε ό,τι αφορά την προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών, να πω ότι ε, πράγματι κάποιοι ε, εξέφρασαν τα παράπονά του ότι είναι πολύ βραχιά η προθεσμία, αλλά ε, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να εκνευρίσω κάποιον από του συναδέλφου. Ε, αυτό δηλαδή οφείλεται στο γεγονός ότι εμείς ως Επιτροπή Πολιτισμού θα πρέπει το νωρίτερο δυνατό να τοποθετηθούμε γιατί έχουμε ακριβώς ειδικό βάρος ως Επιτροπή σε σχέση με αυτό το σύντημα, οπότε θα πρέπει να τοποθετηθούμε από νωρί και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έτσι θέλαμε να δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα από τη δική μας πλευρά. Εάν όμως υπάρχουν τόσοι πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι επιθυμούν να δοθεί λίγο περισσότερος χρόνος για την υποβολή των τροπολογιών, παρότι βέβαια η οδηγία εδώ έχει υποβληθεί εδώ και κάποιες εβδομάδες, εντάξει, σίγουρα να δώσουμε ε, αυτήν την ε, περαιτέρω προθεσμία, δηλαδή να πάει για τις 7 Ιουνίου η προθεσμία ε, υποβολή τροπολογιών, αν πραγματικά τελικά μας βοηθήσει αυτό να έχουμε και ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ε, ε, επειδή όμω εγώ προτείνω πάρα πολλέ διαγραφέ, νομίζω πω ήταν ε, πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Ή κανεί δηλαδή συμφωνεί μαζί μου, είτε ε, δεν συμφωνεί. Και γι' αυτό θεώρησα ότι ήταν εύκολο να θέσω μια τόσο βραχιά προθεσμία. Αλλά εντάξει, υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που επιθυμούν να την παρατείνουμε. Καλώ προτείνω 7 Ιουνίου, λοιπόν, 12 ευρώ το μεσημέρι, ε, ω νέα προθεσμία. Και αν συμφωνούν όλοι, έτσι να το κάνουμε. Έτσι ώστε να έχουν όλοι επαρκή χρόνο στη διάθεσή του για να υποβάλουν τροπολογίε. Ευχαριστώ πολύ. Köszönjük szépen, és akkor a elsőként az árnyék előadók kapnak. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Ας δώσουμε πρώτα το λόγο στους οδησίες εισηγητές και μετά στους συναδέλφους, ε, οι οποίοι μπορούν να μας πούν κατά πόσο θα θελήσουν να παρέμβουν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Πίσας. Εγώ νομίζω ότι η παρουσίαση της οδηγίας για τη βελτίωση της ε, προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών είναι πραγματικά πολύ σημαντική, διότι είναι ένας τρόπος να πούμε στα άνω των 80 εκατομμυρίων ε, ε, πολιτών που έχουν κάποια αναπηρία ότι ε, νοιαζόμαστε για αυτούς. Εάν θέλουμε να έχουμε μια Ευρώπη της ισότητας και της ελευθερίας, είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Εγώ θεωρώ ότι η οδηγία αυτή πρέπει να χρησιμεύσει για να διευκολύνουμε την ένταξη των ατόμων με κάποια αναπηρία στην ε, παιδεία και βελτίωση της ε, πρόσβασης στην αγορά εργασίας μέσω προϊόντων ε, και υπηρεσιών σε ψηφιακό επίπεδο. Πρέπει επίσης να δημιουργήσουμε μια κοινωνία που περιλαμβάνει τους πάντες και να εκμεταλλευτούμε τις νέες τεχνολογίες που έχουμε στη διάθεσή μας προκειμένου να άρουμε οποιοδήποτε εμπόδιο. Με αυτά τα νέα τεχνολογικά μέσα διευκολύνουμε και κάνουμε πιο προσιτή από πλευρά τιμή ε, την πρόσβαση σε αυτά τα προϊόντα και δεν θα πρέπει να χαθεί αυτή η ευκαιρία. Η εξαίρεση των ε, οπτικοακουστικών υπηρεσιών και των ηλεκτρικών ε, ηλεκτρονικών βιβλίων από αυτή την ε, οδηγία ίσως να είναι τεχνικά λογικό, αλλά είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσουμε από πολιτική σκοπιά. Για όλους αυτούς τους λόγους, εμείς από πλευρά της ομάδας μας θεωρούμε ότι είναι αρκετά σημαντικά αυτή η οδηγία, ώστε να ε, δοθεί λίγο περισσότερος χρόνος να την επεξεργασούμε στην Επιτροπή ε, πολιτισμού και ε, θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία Καμέρβερτ να δεχτεί μια πιο ε, μακρά προθεσμία γιατί την περασμένη εβδομάδα λάβαμε τη μετάφραση στις διάφορες γλώσσες και η προθεσμία ολοκληρώνει την Τετάρτη και έχουμε και στη μέση Σαββατοκύριακο. Από πρακτική σκοπιάς δεν υπήρχε χρόνος ούτε για αποφάσεις ούτε για υποβολή τροπολογιών. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι δεδομένη και τις σημασία αυτή τη μεταρρύθμιση, ε, καλό θα ήταν να έχουμε μια νέα ημερομηνία για να καθορίσουμε μια νέα προθεσμία υποβολής τροπολογιών που να είναι λίγο πιο ρεαλιστική, πιο αποτελεσματική και να μπορέσουμε λίγο να ε, επεξεργαστούμε περαιτέρω το θέμα αυτό. Ο κύριος Λόερ, εκ μέρους του κυρίου Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Η Ευρώπη των Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία. Το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Θέλουμε να γίνει και επικύρωση της Σύμβασης του Μαρακέ, που για μας είναι πολύ μεγάλη προτεραιότητα ως πολιτική ομάδα. Βέβαια είμαστε ρεαλιστέ. Η πρόσβαση δεν θα πρέπει να κλείνει πόρτες, ιδιαίτερα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πολλού περιορισμού για την αγαστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και πρέπει να αναζητήσουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση. Η αύξηση της, ε, ε, των δυνατοτήτων της εσωτερικής αγοράς ενδιαφέρει ιδιαίτερα το ECR και το γεγονός ότι κάποιοι θα μπορούν να διαθέτουν στην αγορά προϊόντα ε, ευρύτερα και εκτός συνόρων πρέπει να το αναλύσουμε. Ο κύριος Τζαμπάσκι είναι σκιώδης συγητής για το θέμα αυτό, αλλά ήταν και σκιώδης για το θέμα του UNCRPD, το οποίο υποστηρίξαμε με σθένος. και επομένω θεωρούμε ότι αυτές οι απαιτήσει συνάδουμε με αυτές τις σύμβασεις των ΗΠΑ για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία. Ε, η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή είναι η Επιτροπή ΙΜΚΟ ε, και γιατί αυτή είναι η Επιτροπή που είναι αρμόδια για την εσωτερική αγορά και σε αυτούς επαφίεται να βρουν την κατάλληλη ισορροπία και να υπάρχει πρόσβαση σε αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για όλους, αλλά να μην αυξήσουν και το άχθος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χρειάζεται ενθάρρυνση προκειμένου να υπάρχει συμμόρφωση ε, προς τους κανόνες, αλλά να μην αυξηθεί υπερβολικά το κόστος. Ε, νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια προσέγγιση από την οποία να βγαίνουν όλοι κερδισμένοι και σε αυτή την περίπτωση είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και για την κοινωνία και για τι επιχειρήσει. Επομένω, αυτό μπορούμε να το έχουμε αν έχουμε προϊόντα και υπηρεσίε που είναι προσβάσιμα σε όλου. Από πλευρά ε, τη επιτροπή μα, ε, όπω είπαμε, ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα οπτικοακουστικά μέσα στην πρόταση. Υπάρχουν διατάξει για προσβασιμότητα στην κείμενη οδηγία και θα συζητήσουμε και τη νέα πρόταση σύντομα. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει σαφήνεια και δεν θα υπάρχει καμία έλλειψη ασφάλεια δικαίου για του πολίτε και τι επιχειρήσει και να παρακολουθούμε στενά πώς μπορεί να υπάρχει μια πιθανή σύγκρουση συμφερόντων και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Η παράταση για τις 7 Ιουνίου που πρότεινε η συγγήτρια μας δίνει τη δυνατότητα ίσως να ε, ε, εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε τις κατάλληλες ιδέες και χαιρόμαστε για την πρόταση. Συμφωνούμε. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε. Η ε, κυρία Τρούπελ. ich will auch noch mal και εγώ θα ήθελα ε, να ξεκινήσω κι εγώ με αυτό που αναφέρθηκε, δηλαδή στη διάκριση αφενό σε ό,τι αφορά των προϊόντων που αφορούν τη σύμβαση τη προσβασιμότητα και από την άλλη ε, πλευρά ε, την ανάγκη της, του να επιτύχουμε και να διασφαλίσουμε την επικοινωνία σε ό,τι αφορά τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίε μα. Προφανώ είναι δύσκολο να επιτευχθεί μια ισορροπία εδώ και το βλέπουμε και στην πρόταση τη Επιτροπή, όπου έχοντας εξαιρέσει το σχετικό τομέα από την οδηγία ε, για τα οπτικοακουστικά μέσα. Οπότε, εάν εμεί πραγματικά ε, διαφωνούμε με αυτή την προσέγγιση τη εξαίρεση τη Επιτροπή, θα έχουμε προβλήματα στο να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Υπάρχουν ωστόσο κάποια επιχειρήματα υπέρ του να η, η, τα ζητήματα των οπτικοακουστικών μέσων και τη προβασιμότητά του να ρυθμιστούν στο πλαίσιο τη οδηγία αυτή. Ε, προφανώς και είναι, ε, θα ήταν πιο επιθυμητό να ρυθμιστούμε με τέτοιο τρόπο τα ζητήματα προσβασιμότητας, ούτως ώστε να υπάρχουν περισσότερα ε, άτομα τα οποία θα έχουν πράγματι πρόσβαση, αλλά ε, από την άλλη πλευρά θα πρέπει σε κάθε πλευρά να αποφύγουμε απώλειες ακριβώς επειδή δεν θα υπάρχει κατάλληλη χρηματοδότηση για όλα αυτά. Οπότε είναι περίπληκη η κατάσταση και θα πρέπει να πούμε δηλαδή ότι υπάρχει και το δικαίωμα δε της πολιτισμικής επικοινομορφίας ε, το οποίο είναι και αυτό προς το συμφέρον των ε, καταναλωτών και των χρηστών. Όχι μόνο δηλαδή το ζήτημα της ε, προσβασιμότητας. Οπότε νομίζω Πέτρα μπορούμε να κινηθούμε σε αυτό το πλαίσιο και συμφωνώ και εγώ με την προθεσμία ε, της 7 η Ιουνίου. Ευχαριστώ λέει πρόεδρος κυρία Τινόλφ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τη συνάδελφο την κυρία Κάμερα Βέρτ που πρώτα απ' όλα δέχτηκε να αναβληθεί λίγο η προθεσμία για τις τροπολόγιες στο θέμα της προσβασιμότητας θεμελιώδης δικαιώματων δικαιωμάτων πολιτών πολιτών που ήδη υποφέρουν από δύσκολες συνθήκες και η δουλειά που έχουμε να κάνουμε δεν είναι κάτι απλό. Ώστε να επιτύχουμε κάποια ισορροπία. Υπάρχουν πολλά θετικά σημεία φυσικά, τα οποία ξεχωρίζουν, αλλά είμαι πεπισμένη ότι ζητήματα, όπως ε, αυτό των ε, συστημάτων πρόσβασης της υπηρεσίας, ε, χρειάζεται κάποια εμβάθυνση. Χαίρομαι όμως ε, που αναφερθήκαμε στο θέμα του Μαρακές και είναι ένα ζήτημα σημαντικό την κύρωση της συνθήκης του Μαρακές ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να προβλέψουμε μεγάλη συμμετοχή των ενώσεων για ανάπηρα άτομα για άτομα με αναπηρίες ε, διότι η συμμετοχή τους μέχρι στιγμής υπήρξε περιστασιακή μόνο Τώρα το θέμα της συμμόρφωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών που ουσιαστικά θα γίνεται μέσω της αυτοπιστοποίησης των κατασκευαστών και αυτό χρειάζεται κάποια διαφορετική διατύπωση. Τώρα το θέμα της εφαρμογής της διάταξης της οδηγίας ε, θα πρέπει να αλλάξει κάπως όσον αφορά τον κύκλο ζωής των υπηρεσιών. Ωστόσο είμαι ικανοποιημένη που θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα εμβάθυνσης ε, με αυτή την παραπάνω εβδομάδα που μας προσφέρεται ε, των τροπολογιών γιατί επειδή δεν υπάρχει ακόμα χρονοδιαγράμμα για το ποια θα είναι η επί επιτροπή ε, για αυτή την οδηγία σε κάθε περίπτωση όπως ανέφερε και η συνάδελφος θα προλάβουμε έτσι να παρουσιάσουμε γρήγορα την πρότασή μας πριν από τις άλλες επιτροπές οπότε ούτως ή άλλως ε, θα μπορέσουμε να ακολουθήσουμε την κατεύθυνση της συναδέλφου ωστόσο θα έχουμε περισσότερο χρόνο για να δουλέψουμε στο δεύτερο νομοθετικό θέμα που αφορά την Επιτροπολιτισμού για να δείξουμε ποια είναι η δική μας άποψη. και να ε, έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα εμείς ως Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Φερχάιεν. Ευχαριστώ πολύ ως ε, εισηγήτρια στην ε, επί της ουσίας ε, Επιτροπή ε, θεωρώ πως η σημερινή συζήτηση που γίνεται εδώ είναι πολύ σημαντική και θα συμπεριλάβω αυτά τα επιχειρήματα που αναφέρθηκαν εκεί και στις συζητήσεις στην ΕΜΚΟ. Εκείνο που ανέφερε ήδη η συνάδελφος Πέτρα και το οποίο είχα αναφέρει σε ό,τι αφορά την προσβατισμότητα των ιστοτόπων του δημοσίου τομέα και όπου εκεί είχε προταθεί ε, η συμπερίληψη των σχετικών ε, μέσων, να πω ότι ε, τελικά δεν έγινε αυτή η συμπερίληψη, παρότι είχε αποφασίσει με αυτόν τον τρόπο το Κοινοβούλιο της προηγούμενης βουλευτικής περίοδου, ακριβώς επειδή τώρα με αυτήν την ξεχωριστή οδηγία μπορούμε να επιτύχουμε μια εξειδικευμένη προσέγγιση καλύπτοντας όλον τον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων. Έτσι λοιπόν μπορούμε να έχουμε μια νομοθεσία συνεκτική για ε, όλα αυτά ε, τα ζητήματα. Δηλαδή δεν θεωρώ πως ε, θα πρέπει να έχουμε από τη μία πλευρά σε διαφορετική νομοθεσία να ρυθμίζουμε την προσβασιμότητα των ιστοτόπων του δημοσίου, από την άλλη πλευρά προσβασιμότητα οπτικοακουστικών μέσων του ιδιωτικού τομέα και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, ακριβώς επειδή υπάρχει ήδη τόσο μεγάλη ποικιλομορφία στον, στον σημερινό κλάδο των μέσων ενημέρωση, καλό θα ήταν ε, να προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε αυτά που μα είπε η Πέτρα. Δηλαδή, ε, να εξαιρέσουμε τα σχετικά ζητήματα από αυτή την οδηγία, αλλά δεσμευόμαστε ότι θα υπάρξει μια κατάλληλη ρύθμιση αυτών των ε, ζητημάτων συνεκτικά, ούτως ώστε να μπορέσουμε να, με, με, με, δίκαιο τρόπο να ρυθμίσουμε αυτά τα ζητήματα. Τα τεχνικά ούτως ή άλλως ζητήματα μπορούν να ακολουθήσουν τα όσα θα αποφασιστούν στο πλαίσιο των δύο οδηγιών, που έρχονται και ούτως ή άλλως ε, τα όσα σχολιάζουμε εδώ μπορούν να συμπεριληφθούν στο πλαίσιο τη συζήτηση για την οδηγία AVMS και από εκεί και μετά τεχνικές λεπτομέρειες που θα αποφασιστούν στο πλαίσιο τη AVMS μπορούμε εμεί να τι συμπεριλάβουμε για να ρυθμίσουμε σε ξεχωριστή οδηγία τα ζητήματα των οπτικοακουστικών μέσων. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα των ηλεκτρονικών βιβλίων, νομίζω πω είναι πολύ σημαντικό τόσο οι συσκευέ ανάγνωση, αλλά και οι πλατφόρμε στι οποίε πολλούνται τα e-books να ε, συμπεριληφθούν, να έχουν δηλαδή τέτοιες υποχρεώσεις ε, προσβασιμότητα. Ε, τώρα τα ηλεκτρονικά βιβλία τα ίδια θα πρέπει να, είναι, να, να παράγονται σε τέτοιο, να διατίθενται σε τέτοιο μορφότυπο ώστε να είναι αναγνώσιμος αυτό ο μορφότυπο από τις σχετικέ συσκευές, τις προσβάσιμες συσκευές ανάγνωση Οπότε ε, αυτό το ζήτημα βέβαια ε, θέτει το ερώτημα του κατά πόσο θα ε, αποκλειστούν εντελώ από το βιβλίο εφαρμογή στα ηλεκτρονικά βιβλία ή κατά πόσο ξεχωρίζουμε το περιεχόμενο, δηλαδή τα ίδια τα books, από τι συσκευέ μέσω των οποίων καθίσταται διαθέσιμε και οι πλατφόρμε μέσω των οποίων πολλούνται τα ηλεκτρονικά βιβλία. Η συνάδελφο Καμπέβεται ούτω ή άλλω κάνει αυτό το διαχωρισμό μεταξύ δηλαδή του περιεχομένου των βιβλίων και των συσκευών ανάγνωσή του και βλέπουμε ότι αντίστοιχη προσέγγιση ακολουθούνται για παράδειγμα και στον εθνοτικό τομέα σε βιβλιοθήκες ή σε άλλες, ή άλλους τέτοιους ε, βιβλιοθήκες σε μικρότερες, ε, μικρότερου μεγέθους όπου ακριβώς υπάρχουν και τέτοιου είδους απαιτήσει προσβασιμότητας. Οπότε μπορούμε να επιτύχουμε τον ελάχιστο κοινό παραδομαστή. Τώρα, ε, κάτι το οποίο ακόμα θα πρέπει να γνωρίζουμε σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση, αξιολόγηση αντικτύπου για την προσβασιμότητα που θα γίνει από την πλευρά της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς. Να πούμε ότι οι αριθμοί ε, που θα υποβληθούν εδώ είναι από το 2011-2012, οπότε είναι λίγο παροχημένοι αυτά οι αριθμοί. Ε, και άλλωστε το 2012 υπήρξε συμφωνία μεταξύ των Υπουργών σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα, ότι δηλαδή θα πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα. Μέσα στα τελευταία λοιπόν 3-4 χρόνια ακριβώς λόγω αυτής το πρωτοβουλία, μέσω των λέω, τεχνικών καινοτομιών που κατέστησαν ε, με δυνατές και μέσω των, ε, του διαδικτύου έχουν αλλάξει πολλά. Οπότε εγώ ασκώται κάποια κριτική στα απορίσματα της αξιολόγησης αντικτύπου ακριβώς γιατί δεν απηχεί αυτή η αξιολόγηση αντικτύπου τη σημερινή κατάσταση όπως έχει. Ε, ε αναφέρεται δηλαδή σε μια περίοδο που δεν είχαν γίνει τόσα όσα έχουν γίνει σήμερα. ε, ε Άλγα Τρούπελ και η Πέτρα Κάμα έβατε, το ανέφεραν ήδη ότι ενδεχομένω να μην γίνεται κανεί πολύ δημοφιλή όταν αναφέρεται σε κάτι τέτοιο. Αλλά ε, σίγουρα γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να λάβει υπόψη το ε, ποιε εξειδικευμένε απαιτήσει θα ισχύουν για παράδειγμα μικρότερε επιχειρήσει ή για οντότητε ε, οι οποίε περιλαμβάνουν τέτοιου είδου οπτικοακουστικά μέσα. Δηλαδή, τι είδου υποχρεώσει επιβάλλω σε όλου αυτού του φορεί και τι επιτυχάνω τελικά στην πράξη και ε, στο πλαίσιο της ε, προσβασιμότητας των ε, δημόσιων ιστοτόπων είχε αναφερθεί αυτό, δηλαδή όλο αυτό το επιπρόσθετο άχθος το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις είναι, δεν είναι απαραίτητο, δηλαδή θα πρέπει να ληφθεί και αυτό το ζήτημα υπόψη όταν συζητάμε τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία και τη σχετική προσβασιμότητα. Δηλαδή, δεν προστατεύουμε με αυτόν τον τρόπο τα δικαιώματα του, εάν τελικά προβλέψουμε ένα τόσο περιοριστικό κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο τελικά να μην επιτρέπει τόσο πολύ διαθέσιμο υλικό τελικά, τόσο πολύ διαθέσιμο περιεχόμενο και για τα άτομα με την αναπηρία, ακριβώς επειδή προβλέπουμε τέτοιου είδους περιοριστικούς κανόνες για όλα όσα ε, προσφέρονται στην αγορά. Δηλαδή τελικά θα έχουμε επιτύχει ένα ε, ίσους περιορισμούς για όλους, αλλά τελικά δεν θα είναι προς όφελος αυτό τελικά όλων μας. Ευχαριστούμε πολύ. Κάποιος άλλος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να παρέμβει για το σημείο αυτό. Όχι. Να ξαναδώσουμε λοιπόν το λόγο στην εισηγήτρια. Παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ τους συναδέλφους για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα ήθελα να κάνω δύο ακόμα παρατηρήσεις. Νομίζω πως ως Επιτροπή Πολιτισμού θα πρέπει να περιοριστούμε στα όσα εμπίπτουν στο δικό μας τομέα αρμοδιότητες, δηλαδή ε, υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και ηλεκτρονικά βιβλία. Δεν νομίζω πως θα έπρεπε εμείς τώρα να δώσουμε συστάσεις στην Επιτροπή ΙΜΚΟ για όλα ε, τα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία ε, καλύπτει αυτή η πράξη προσβασιμότητα. Δηλαδή το να προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε τη γνώμη σα στην ΙΜΚΟ δεν είναι κάτι το οποίο θα μα εξυπηρετούσε. Ειδικότερα όταν θα ε, πιστεύουμε και στη σχετική συζήτηση με την ΙΜΚΟ επί των λεπτομεριών. Και για να είμαι σαφής, να επαναλάβω ότι προφανώ επιθυμώ περισσότερη προσβασιμότητα στο πλαίσιο των οπτικοακουστικών ε, μέσων και των σχετικών υπηρεσιών και ηλεκτρονικών βιβλίων για άτομα με αναπηρία, ε, με βαρικοία και ούτω καθεξής. Αλλά αυτό που λέω είναι ότι θα πρέπει να επιτύχουμε την κατάλληλη ισορροπία. Και φυσικά αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι δύσκολο να το περάσουμε ως μήνυμα, γιατί εύκολα δηλαδή μπορεί να κανείς να εκτεθεί στον κίνδυνο του να τον κατηγορήσουν ε, ότι η Επιτροπή Πολιτισμού δεν θέλει να κάνει τίποτα για τα άτομα με αναπηρία, δεν θέλει να τα προστατεύσει. και αυτό το είπε ε, και μόλι τώρα και η Ζαμπίνε. Εκείνο που θέλουμε να εξασφαλίσουμε από τη μία πλευρά να συνεχίσει να υπάρχει ποικιλομορφία, να υπάρχει μια μεγάλη προσφορά ε, και από την άλλη πλευρά να διασφαλίσουμε και την κατάλληλη προσβασιμότητα. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να δούμε πόσο μπορούμε να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία και θα πρέπει να αναζητήσουμε ποιοι είναι εκείνοι με τους οποίους θα επικοινωνήσουμε τόσο ώστε να έχουμε να γίνουν οι να επιτύχουμε τις κατάλληλες συμφωνίες έτσι ώστε να διασφαλίσουμε περισσότερη προσβασιμότητα στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών ε, μέσων και ηλεκτρονικών και στα ηλεκτρονικά ε, βιβλία. Και αυτό σημαίνει βέβαια ότι χρειάζεται μια ξεχωριστή οδηγία, ε, μια ξεχωριστή νομοθετική πράξη σε αυτά τα ζητήματα. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε και σχετικές προτάσεις σε ό,τι αφορά την οδηγία AVMS. Ε, γνωρίζω πως ένα ακόμα πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν ισχυρές αντιστάσεις στο επίπεδο του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά αυτήν την πρόταση, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα, τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, αλλά και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον περιοριστικό χαρακτήρα τελικά όλης αυτής της πρότασης και το τι θα μπορούσε να, να, να σημαίνει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν να συνεχίσουμε εμείς τις δικές μας ε, ε, προσπάθειες σε σχέση με μια ξεχωριστή δουλειά από το να περιμένουμε, αντί να περιμένουμε το τι ακριβώς θα γίνει και πότε τελικά θα συμφωνηθεί αυτή η οδηγία EVMS και πότε θα μπορέσει να περάσει και από το Συμβούλιο. Άρα λοιπόν νομίζω πως ε, ε, καλύτερο θα ήταν να, ε, με την ξεχωριστή οδηγία να νομίζω ότι θα μπορούσαμε να επιτύχουμε ταχύτερα αποτελέσματα από, ό,τι, από την οδηγία που πρότεινε μόλις τώρα η Επιτροπή. Και Ήδη έχω διαβάσει διάφορε γνωμοδοτήσει από εκπροσώπου κυβερνήσεων και είδα ότι και εκεί δεν υπάρχουν τόσο πολλέ θετικέ αντιδράσει απέναντι στην προτινόμενη οδηγία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, για να συνοψίσουμε, συμφωνούμε με τη νέα προθεσμία υποβολή τροπολογιών 7 Ιουνίου στις 3 το μεσημέρι. Και τώρα στις 13 Ιουλίου θα έχουμε την ψηφοφορία στην Επιτροπή Πολιτισμού. Εδώ μπορούμε να κλείσουμε το σημείο αυτό. Θα τα ξαναπούμε στις 20 Ιουνίου του 2016 από τις 3 μέχρι τις 6.30 το απόγευμα και 21 Ιουνίου από 9 μέχρι 12.30 και από 3 μέχρι 6.30. Η Πρόεδρος ε, πολύ ευγενικά ευχαριστεί και τους Δερμηνείς και τη Γραμματεία. Το δημόσιο λοιπόν κομμάτι της συνεδρίασης κλείνει και σε λίγο θα ακολουθήσει η συνεδρίαση των συντονιστών. Ευχαριστώ.